Καλησπέρα συνάδελφοι. Να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Είμαστε στο σημείο 13 της ημερήσιας διδαξής μας, όπου πρέπει να ψηφίσουμε τα τρία σχέδια έκθεσης, την απαλλαγή για τις τρεις αρχές Παρακαλώ δοκιμάστε τις ε, κάρτες σας και ξεκινάμε με έναν έλεγχο. Κάνουμε πρώτα ένα τεστ. Ο κύριος Λούντβικσον. Θα προβλέψουμε πρόστιμα. Without flexibility. Χωρίς καμία ευελιξία. Ωραία. Εψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Put the voting camera are not voting. Can everybody vote, please? Δύο βλέπω δεν έχουν ψηφίσει. Ψηφίστε. Εντάξει δεν είναι και υποχρεωτικό. Πρώτα. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Απαλλαγή. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμ... Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε άρχεται. Vote is closed. Πέρας. Μία ψήφος κατά μόνο και τέσσερις αποχές εγκρίνεται. ΕΙΟΠΑ. Συμβαστική Α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται, συγγνώμη. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο που τροποποιήθηκε έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 41 υπέρ, ένα κατά, 4 αποχέ. Εγκρίνεται. Έσμα τώρα. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο που τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, 41 υπέρ, μία, ένας κατά, τέσσερις εποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στο σημείο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 Uh, Όπως ξέρετε, έχουμε ένα πολύ σημαντικό τραπεζικό πακέτο, το οποίο συναποτελείται από μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες τροποποιούν το CRR, το CRD και το BRD. Έχουμε διαιρέσει σε δύο διπλωματικέ ομάδε το σύνολο αυτών των κειμένων. Το ένα για το CRR και το CRD, με επικεφαλή τον κύριο Ζήμων. Και το άλλο, του οποίου ηγείται ο κύριος Χόκμαρκ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι τομείς επικάλυψης μεταξύ των δύο. Διότι όπως τα γνωρίζετε, οι διατάξεις του CRR-CRD ε, μπορεί να είναι διαφορετικές από το άλλο σκέλος του πακέτου, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζουν. Δεν είναι ακριβώς ε, θέμα επικάλυψης. Είναι αλληλένδετοι τομείς σε πολλές περιπτώσεις, αν και το CRR-CRD καλύπτουν πολύ περισσότερα θέματα. Όμω στο δεύτερο σκέλο υπάρχει και μια ξεχωριστή νομοθετική πρόταση, η οποία αφορά και τον BRD, αλλά κυρίω έχει την ιδιαιτερότητα να αναφέρεται στο subordination. Για να τα κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο περίπλοκα, στην πρώτη ομάδα ξέρουμε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ πιεστικά για την υλοποίηση και ίσως να χρειαστεί και ταχεία διαδικασία για ένα κομμάτι του CRD, CRD, CRR. Για το IFRS 9. Έχουμε επίσης δύο σημεία. Το, ε, τα διεθνή πρότυπα 9 και το και την υπόταξη που μπορεί να χρειαστεί να περάσουν από την ταχεία διαδικασία επίσης. Ε, παράλληλα, σήμερα θα προχωρήσουμε με χρονική σειρά τις δύο εκθέσεις, στην εξέταση των δύο εκθέσεων. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντοτε αυτά αποτελούν πακέτο και μπορούμε να αποφασίσουμε να προχωρήσουμε διαφορετικά. Αν θέλουμε να ακούσουμε τους δύο, σκιο, τους δύο εισηγητές και τους σκιώδεις, να έχουμε και γενική συζήτηση, ίσως για αυτή την πρώτη φορά για σκοπούς ε, σαφήνειας να ακολουθήσουμε την ε, γραμμική πορεία, αλλά να θυμόμαστε ότι αυτά πάνε παράλληλα. σε μια οργανωμένη κοινή ομάδα, ιδίως στις περιοχές όπου υπάρχει η, επαφή, η κοινή επαφή. Να δώσω τώρα το λόγο στον Γκούναρ Χόκμαρκ, ο οποίος είναι εισηγητής του πρώτου πακέτου. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την ευθύνη αυτή με αυτό το ζήτημα. Έχουμε την οδηγία για την ε, καθάριση των τραπεζών και τις νέες προτάσεις. Και όπως είπατε και εσείς υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες συνδέσεις ε, με το τμήμα CRR. Αυτό, όπως είπατε και εσείς, είναι φυσιολογικό και γιατί υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο, αλλά και γιατί ουσιαστικά είναι δίδυμα παιδιά. Γεννήθηκαν την ίδια στιγμή, μετά την κρίση. Θέλαμε λοιπόν με την νομοθεσία να έχουμε τις ε, κεφαλικές απαιτήσεις αλλά και ταυτόχρονα στην αγορά κανένας να μην θεωρεί να ε, δρά ε, με την πεποίθηση ότι θα τον διασώσουν. Εγώ ανέλαβα τον BRRD. Συνεργαστήκαμε, πολύ καλή δουλειά κάνουμε. Το έχω πει όμως της συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας ότι πρόκειται για ένα είδος αναζωογόνηση του καπιταλισμού στη χαρτοπιστωτική αγορά. Και είδα ότι είναι κάτι που υποστηρίζεται τελικά. Οι τραπεζίτες ε, παίρνουν το μερίδιο, τη μερίδα του λέοντος της ευθύνης όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε τώρα λοιπόν την ε, νομοθεσία τη σχετική λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, φρέσκα πράγματα, φρέσκο πράγμα μάλλον και Πολλοί τώρα προσπαθούν να δουν στην πράξη πώς όλα αυτά θα λειτουργήσουν. Παρακάμπτεται η οδηγία, δεν χρησιμοποιείται όσο πρέπει. Εγώ διαφωνώ και θεωρώ ότι αρχές και κυβερνήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν νέα τραπεζικά προβλήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται στους κανόνες και να τους ε, τηρούν. Και πάντα βέβαια εφαρμόζοντας την νομοθεσία, γιατί αλλιώς θα βλέπαμε πολλά προβλήματα, όπως τα είδαμε και με τον παραδοσιακό τρόπο αντιμετώπισης των τραπεζικών προβλημάτων μέχρι τώρα. Ποια θα ήταν τα αρνητικά όμως αποτελέσματα. Πρώτον, ότι θα υπονομευόταν περισσότερο ακόμη η δημοσιονομική σταθερότητα και τα δημοσιοοικονομικά των κρατών μελών, αλλά δεν είναι αυτή η μόνη συνέπεια. Αν στέλναμε τελείω ασφαλμένα μηνύματα στι αγορέ. θα είχαμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί το λέω αυτό. Όταν θεσπίστηκε η οδηγία BRRD, ουσιαστικά πρόκειται για δύο σημαντικούς στόχους που υπηρετούσε αυτή η οδηγία. Ο ένας στόχος ήταν όταν μια τράπεζα εκαθαρίζεται, θα πρέπει ε, να γίνεται γρήγορα, με το σωστό τρόπο, με διαφανή τρόπο, να ακολουθούνται ήδη οι κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην διασώζονται από τα κράτη τράπεζες. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος και ο δεύτερος στόχος ήταν να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στις αγορές ότι τώρα υπάρχει ένα νέο καθεστώς. Και από αυτήν την έννοια η οδηγία BRRD έχει δύο, σημαντικούς, δύο σημαντικά καθήκοντα. Πρώτον, αν έχουμε ανάγκη καθάριση μιας τράπεζας, θα πρέπει να ξέρει κανείς πώς θα το κάνει αυτό και θα πρέπει να γίνει με ίδια κεφάλαια. Το άλλο όμως θέμα είναι η κίνδυνη για τις τράπεζες που εισέρχονται σε διαδικασία καθάρισης, αν λειτουργεί οδηγία, θα είναι πολύ λιγότερη κίνδυνη. Γιατί ανάλογα θα βαθμολογούνται από τις οικοσαξιολόγησεις οι τράπεζες, ανάλογα με τους κινδύνους, με τα ρίσκα. Έχουμε λοιπόν αυτό το πακέτο εδώ για, το, για την οδηγία BRRD. Είναι ένα πολύπλοκο πακέτο. Έχει να κάνει με το πώς θα προσαρμοστεί η οδηγία στις νέες εξελίξεις, για παράδειγμα στο TILAC και τα MREL. Τη διαθεσιμότητα, μάλλον την ελάχιστη απέτηση δύο κεφαλών επιλέξιμων υποχρεώσεων. Και νομίζω ότι ένα από τα θέματα που τα συζητούσαμε τότε, όταν δηλαδή ξεκινήσαμε με την οδηγία BRRD ήταν ότι δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια αυταπάτη, ότι δηλαδή μόνο ένα μέρος του κεφάλαιου των τραπεζών είναι εκτεθειμένο, αλλά θέλαμε να υπάρχει μια μεγάλη ομοιότητα των τραπεζών και με άλλες επιχειρήσεις, ότι δηλαδή όλο το κεφάλαιο είναι σε κίνδυνο αν κάτι δεν πάει καλά, όχι μόνο ένα τμήμα του. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί Τότε λέγαμε ότι θα έχουμε συγκεκριμένα τμήματα του κεφαλαίου που θα πηγαίνουν για τη διάσωση με ίδια μέσα. Όμως υπήρξε ευρύτατη συμφωνία ότι αυτό θα αποδυνάμουνε το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της BRRD και θα δημιουργούσε προβλήματα για την αναχρηματοδότηση αυτών των τμήματων του κεφαλαίου. Γιατί αν μπαίνει σε κρίση σιγά σιγά μια τράπεζα, είτε θα ε, ήταν πολύ ψηλά τα επιτόκια, είτε πολύ λίγοι θα συνεισέφεραν αν ήξεραν ότι ακριβώς αυτό είναι το συγκεκριμένο κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση με ίδια μέσα και αν πρέπει να πάρει ένα σημαντικό δάνειο αυτή η τράπεζα. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι η συζήτηση για την υπαγωγή αυτή, για την ε, υπόταξη, είναι κάτι σημαντικό. Το θέμα όμως είναι να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και νομίζω ότι το υπηρετεί αυτό η παγωγή. Και βέβαια ε, και την πιο ε, γρήγορη εκαθάριση υπηρετεί ως στόχο. Αλλά είναι σωστό να το κάνουμε σωστά. Είναι σημαντικό μόνο να το κάνουμε σωστά, γιατί τελικά βλέπουμε ένα χρόνο μετά την εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος να δημιουργείται ένα πρόβλημα που θέλαμε να αποφύγουμε όταν ε, θεσπίσαμε αυτό το νομοθέτημα. Πρέπει να δούμε λοιπόν την ευρύτερη προοπτική της νομοθεσίας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν ίσως πιο σκόπιμο και αυτό το τμήμα του πακέτου να ενταχθεί στα άλλα δύο. I think we all have discussed Είμαστε ανοιχτοί βέβαια. Εγώ και όσοι έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να αποφύγουμε να κάνουμε κάτι λάθος. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια ενοποίηση με τα περί BRRD στο όλο αυτό πακέτο. Σε ό,τι αφορά το TILAC, τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Θα εφαρμόζεται, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, μόνο στις μεγάλες ε, και σημαντικές αποσυστημικές πλευράς τράπεζες θα πρέπει να δούμε και τον ηθικό και το τίλακ, οι μεγάλες τράπεζες. Να μην έχουμε μεγαλύτερα κεφάλαια από αυτά που χρειάζονται. Γιατί πάλι το παραλαμβάνω. Αν δυσκολεύονται τράπεζες να δανείζονται, να δανείζουν, συγγνώμη, επανερχόμεθα στην κατάσταση που δημιούργησε την ε, δημοσιονομική αστάθεια, ότι οι εταιρείε ε, δεν μπορούσαν να πάρουν ε, δάνεια, πάχουσαν οι αγορές, υπήρξε πολύ ανταγωνιστικότητα. Άρα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αφενό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και αυτών των ευκαιριών τράπεζε να χρηματοδοτούν τι απαιτούμενε επενδύσει. Ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να έχουμε τον ίδιο ρυθμό και με τα άλλα σκέλη του πακέτου να κινούμαστε παράλληλα. Θα το συζητήσω με τον ε, Πέτερ Σίμων. Θα δούμε και με τους σκιώδεις λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ένα είδους παραλληλισμού ευθυγράμμισης πρέπει να υπάρχει. Αυτό το πακέτο σίγουρα είναι λιγότερο πολύπλοκο σε σχέση με το CRR. Ίσως μπορεί να, έχει, ε, να πάμε λίγο ένα βήμα εμείς πιο μπροστά για να διασταυρώνουμε τις ε, αναφορές, αλλά Επειδή κλείγει ο χρόνος μου τώρα, έχω 30 δευτερόλεπτα, στα 10 λεπτά που μου δώσατε, σας τα γυρίζω πίσω τα 30 δευτερόλεπτα. Πρόεδρος, μήπως θα τα χρησιμοποιήσετε για να απαντήσετε στο ερώτημα, αν θεωρείτε σκόπιμο να έχουμε μια ταχεία διαδικασία για την υπαγωγή. Απάντηση. θα πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν θέλω να έχουμε την υπαγωγή στην βαθμολόγηση του χρέους και μετά να έχουμε τη συζήτηση ειδικών τμήματων ε, του κεφαλαίου για τον Μπέιλιν και να τα ξανασυζητήσουμε. Εγώ νομίζω πρέπει να επιλέξουμε όλο το κεφάλι. Ένα πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι κάποιοι πίστεψαν ότι δεν θα χρησιμοποιείται αυτό το κεφάλαιο για τη διάσωση. Πρέπει ξεκαθαρίσουμε από την αρχή αυτά. Ε, Πέτρο Σίλβα Περέιρα. Πέτρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αναθεώρηση των ε, κανόνων τραπεζικής διοργάνωσης πρέπει να βασιστούν στο πλαίσιο που μας προτείνει και ο εισηγητής, ο κύριος Εκμαρκ. Δηλαδή να αποτιμήσουμε τους πρόσφατους και ισχύοντες κανόνες, αλλά να δούμε και την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τώρα ε, για να κάνουμε τη σχετική αξιολόγηση. Και όσο και αναλυθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ε, υποβάλλει ένα πακέτο προτάσεων, είναι επειδή αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια σειρά προβλημάτων που πρέπει να επιληθούν. Πέρα από την απαραίτητη προσαρμογή στα καινούργια διεθνή πρότυπα, τα οποία μας δεσμεύουν. Θεωρούμε ότι αυτή η δέσμη μέτρων της Επιτροπής Ιδίω ό,τι αφορά τους κανόνες ρύθμιση. Και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών είναι θετική κίνηση και πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αντιμετώπισης των ε, αντικσότητων και των διαφόρων ε, κλειδονισμών του συστήματος και για να έχουμε πιο ομοιόμορφο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάμε λοιπόν στη σωστή κατεύθυνση για να εμβαθύνουμε την τραπεζική μας ένωση. Πέραν αυτών, όπως είπα και προηγουμένως, η ανάγκη να προσαρμοστούν αυτοί οι κανόνες στα διεθνή πρότυπα είναι κάτι το πραγματικό, όπως και το γεγονό ότι να λάβουμε υπόψη τη ιδιαιτερότητε του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματο όμω. Και τις διαφορές που εντοπίζουμε στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Εκεί απαιτείται κάποιο περιθώριο ευελιξίας, κάποια διαλλακτικότητα στην ε, ρύθμιση. Η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος είναι κάτι που πρέπει να το επιδιώξουμε με τρόπο ευφύ, χωρίς να υπονομεύσουμε τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία. Δεν θέλουμε να θέσουμε τέτοια επίπεδα απαιτήσεων που να οδηγήσει σε στη δημιουργία ενός τέτοιου βάρους που θα είναι επιζήμιο για τον τελικό μας σκοπό που είναι η ανάπτυξη, η περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. Ε, ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, διασφαλίσεις, κάποιες δεκλίδες ασφαλείας, καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης αυτών των κανόνων. Σε πρώτη φάση, σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση της ιεραρχίας των πιστωτών, βλέπουμε ως θετικό σενάριο την δυνατότητα να αυτονομηθεί η πρόταση αυτή. Και να υπάρξει μια ταχεία εναρμόνιση, αλλά ταχύτερο θα πρέπει να είναι ε, το πέρασμα στην αγορά. Για την νέα κατηγορία «χρέος» που προτείνεται και που δεν θα υπάρχει η προτιμησιακή μεταχείριση. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες Μορέλ, πρέπει να υπάρξει ο συντονισμός ε, των ευρωπαϊκών κανόνων βάσει των όσων προβλέπει το Βερολίνο και τα διεθνή πρότυπα στο πλαίσιο του ΤΙΛΑΓ. Αυτός ο συντονισμός είναι ένα από τα θετικά στοιχεία του πακέτου προτάσεων της Επιτροπής και θα επιτρέψει τη μείωση του και τον περιορισμό του κατακαιρματισμού των κανόνων. Σε κάθε περίπτωση επιμένω. Το επίπεδο απαιτήσεων πρέπει να είναι λογικό. Πρέπει να είναι ε, ανάλογο με τις ε, διαφορετικές καταστάσεις, με την ποικιλία τους. Είναι λογικό οι τράπεζες συνολικής συστημικής σημασίας να υπόκειται σε ιδιαίτερους κανόνες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και τέλος, πρέπει προφανώς να περιορίσουμε στο ελάχιστο το κόστος. Το κόστος που θα επιφέρουν οι νέες αυτές απαιτήσει. Για τον τραπεζικό κλάδο, πέραν της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μέσω των πιστώσεων. Τέλος, ήθελα να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα προβλήματα. Το πρώτο, έχει να κάνει με τη διάρθρωση των κανόνων στο λεγόμενο στην ελαχιστοποίηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων στο MRL e και στο Bailin, τη διάσωση με ίδια μέσα, και ε, την ε, κάλυψη των καταστάσεων όπου εμπλέκονται για τρίτα κράτη. Σε δεύτερη φάση, η σημασία της θέσπισης νέων κανόνων, που είναι και ένα μεταβατικό σύστημα και το οποίο θα διασφαλίζει την προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο θα επιτρέπει συγκεκριμένα να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα κάποιων ιδιαίτερων κατηγοριών χρέους, τα οποία είναι εκτός βάση των ισχυόντων κανόνων. Αυτά θέλαμε να επισημάνουμε στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και εντός ενός επικοδομητικού διαλόγου που ελπίζουμε ότι θα κατατήσει ο συνάδελφος ε, Χόκμαρκ. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα επόμενα βήματα. Uh, e Ευχαριστώ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Δεν βλέπω τον κύριο Καμάλ. Κάποιος που θέλει να διαβάσει εκ μέρους του. Εγώ είμαι εδώ για το CRD4 και CCR2. Α, δεν είμαι για αυτό ακόμα. Εντάξει, θα περιμένω. Ναι, θα περιμένετε αν δεν έχετε συγκεκριμένα κάτι να μας πείτε για αυτό το θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας δώσω μετά το λόγο όταν περάσουμε στην έκθεση Ζήμων. Mm. Η Σιλβί Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γκούναρ, να είμαστε πάλι εσείς και κάποιοι άλλοι ακόμη για αυτό το νέο πακέτο. Να επαναλάβω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο Γκούναρ. Τα σχόλια που ακούγονται για την εφαρμογή των κανόνων ε, που εφαρμόσαμε στην προηγούμενη εντολή. Εδώ περάσαμε από το Βερολίνο στους νέους κανόνες, δεν είναι απλό και σε αυτό το πλαίσιο νομίζαμε ότι θα υπάρχουν κάποιες άλλες δυνατότητες εξαίρεσης, κάτι που δεν ήταν και ένα δίκο. Απλώς να σας πω ότι προσυπογράφω σε αυτή την προσέγγιση που είναι πραγματιστική, πραγματιστική και στη συνέχεια όσων έχουν ήδη γίνει. Επίση, γι' αυτό που υπόθηκε περί κατακαιρματισμού το θεωρώ σημαντικό, διότι σε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει στην Τραπεζική Ένωση, ε, συνειδητοποιούμε ότι ένα στόχο που θα πρέπει να έχουμε και αυτό αφορά όλα τα κείμενα που έχουμε μπροστά μα είναι να καταπολεμήσουμε τον επανακαιρματισμό τη αγορά και να βεβαιωθούμε ότι θα κυκλοφορούν και πάλι κεφάλαια ε, ανεμπόδιστα και διασυνοριακά. Αυτό αναζητούμε στην ενιαία αγορά. Επίση, κατά την άποψή μου, δείχνει ότι η συνείδηση μεταβάλλεται περί των θεμάτων αυτών. Και τελευταίο σημείο που είναι σημαντικό για μένα να έχουμε κατά νου την ανάγκη να υπάρχουν ισότιμοι κανόνε παιχνιδιού βάσει της Βασιλείας. Δηλαδή να ξέρουμε πώς διοργανώνουμε την όλη συζήτηση. Θέλουμε να είμαστε πιο διαφανεί με περισσότερη λογοδοσία σίγουρα, αλλά θέλουμε να μπορούμε να τηρούμε για κάποιες υποσχέσει και να τιμούμε και τους εταίρους μα που τι τηρούν επίση, Με τι αβεβαιότητε των Ηνωμένων Πολιτών αυτή τη στιγμή ανησυχούμε και είναι λογικό. Ε, οπότε σε αυτό το συνολικό πλαίσιο πρέπει να δούμε τα κείμενα αυτά υπό τη συγκεκριμένη οπτική γωνία και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσουμε να συνεργαστούμε και πάλι και θα ήθελα να ορίσουμε ένα ρυθμό εργασία αρκετά ε, ταχύ. Ε, πραγματικά εκπλήσωμαι που βλέπω ότι ο ρυθμός εργασίας της Επιτροπής ΑΕΚΟΝ σε αυτή τη θητεία έχει λίγο επιβραδυνθεί σε σχέση με την προηγούμενη θητεία. Αυτό λιγάκι θα γυρίσει μπούμερα για να μπει φοβάμαι. Ευχαριστώ. Βλέπω τον κύριο Καμάλ που ήρθε. Οπότε είστε έτοιμος να σας δώσω τον λόγο. Ε, εκτός αν θέλετε να περιμένετε λίγο. Ναι, μπορώ, μπορώ να περιμένω, λέει ο κύριος Καμάλ. Ωραία, λοιπόν. Φάμπιο Ντεμάζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με χαρά συνεργάζομαι και πάλι με τον Γκίνορ Δεν έχουμε τελειώσει βεβαίω λοιπόν ακόμα. Ελπίζω να είμαστε κάπως πιο παραγωγικοί. Πριν μπούμε στην συζήτηση να πω ότι διαφωνώ με κάτι το οποίο ακούω ξανά και ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχουμε δηλαδή κάποια υπερβολική ρύθμιση που θα αποτελέσει εμπόδιο στο να παρέχουν οι τράπεζες πίεση στην πραγματική οικονομία. Δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα για κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι στις ΙΠΑ ε, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, αλλά ε, ήταν ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα στο Ντόντ Frank. Είχαμε τους ίδιους κανονισμούς σε διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, πολιτική δανεισμό. Οπότε το βασικό εμπόδιο για το οποίο δεν δανείζουν τράπεζες είναι ότι έχουν πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα για την κερδοσκοπία που έκαναν προκρίσεις. Δεν έχουν επιλύσει το θέμα των κακών στοιχείων που έχουν στον ισολογισμό τους και δεν υπάρχει και ζήτηση στην αγορά. κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν και οι εμπειρικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε οι περισσότεροι δεν θα έλεγαν ότι η ρευστότητα είναι το βασικό πρόβλημα, αλλά μάλλον η ζήτηση και γι' αυτό δεν υπάρχει αρκετή παροχή πίστης. Οπότε, καλό είναι να συμφωνήσουμε σε αυτή την αφετηρία και να μην προσπαθούμε συνεχώς να νερώσουμε τους κανόνες. Για μας έχει σημασία λοιπόν να έχουμε ένα αξιόπιστο Μπέιλιν ε, και μετά θα προχωρήσουμε στην ίδια την ε, αναδιοργάνωση των τροπεζών. Να αναφέρω λοιπόν τώρα τρία σημεία. Θεωρούμε ότι οι βασικές παγκόσμιες προδιαγραφές ε, για τη συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών έχουν ενσωματωθεί και αυτό αφορά τις 13 παγκόσμια σημαντικές συστημικές τράπεζες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιπε τράπεζε όμως που είναι υπό την άμεση υποπτία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να συμμορφωθούν μόνο με το Ευρωπαϊκό Εμπρέλ, την ελάχιστη απέτηση δύο κεφαλαίων ε, και επιλέξιμων κεφαλαίων που είναι πιο ε, ελαστικό καθεστώ. Και βεβαίω, ε, το μεγαλύτερο κομμάτι των αποφάσεων βρίσκεται στα χέρια των αρχών διάσωσης. Επίσης υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες ε, δομημένες ε, ε, κάποια στοιχεία και θα κρίνουν οι αρχές διάσωσης κατά περίπτωση και δεν υπάρχει μια ιεραρχία των πιστωτών. Αυτό δημιουργεί λοιπόν περισσότερη αβεβαιότητα και όχι περισσότερη σαφήνεια και γίνονται πιο περίπλοκοι Και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θέλει να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία επιλέξιμη για Μπέιλιν και γνωρίζουμε πως υπάρχουν τέτοια μέσα. Υπάρχουν οι κανόνες ε, για το κεφάλαιο Tier 1 και Tier 2 και ότι Όφελο και αν προσδοκούν οι τράπεζε από αυτέ τι κατηγορίε, θεωρούμε ότι θα είναι ει βάρο της βεβαιότητας και τη αφήνεια και δεν θα γίνει έτσι το εργαλείο απλούστερο και πιο αξιόπιστο. Θεωρώ λοιπόν πω έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συζητούνται με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και για λόγου αναλογικότητα και εξαίρεση μικρότερων χρηματοπιστωτικών δρυμάτων, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. σύντομα. πολλά υπόθηκαν. Θα ήθελα να πω επίσης πως ο τόνος της συζήτησης έχει σημασία και θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία όταν θα μιλάμε για το CRD και CRR, τις οδηγίες κεφαλαιακών απαιτήσεων. Έχω και εγώ τις ίδιες παρατηρήσεις με αυτές που έκανε ο Φάμπιο, ότι υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει να διαλέξουμε, δηλαδή ότι είτε θα έχουμε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, είτε στη βαρύ ρύθμιση των τραπεζών και ότι η διαθέσιμότητα πίστοση σχετίζεται με τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα για κάτι τέτοιο. Ίσως βραχυπρόθεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς οι αυξήσεις του κεφαλαίου, κεφαλαίου θα εισαχθούν γρήγορα ή αργά ή σε ποια στιγμή του επιχειρηματικού κύκλου, αλλά δεν σημαίνει ότι θα επιλέξουμε το ένα ή το άλλο. Το αντίστροφο ισχύει. Μόνο οι τράπεζες που έχουν επαρκή κεφάλαια μπορούν να αναλάβουν κινδύνους και μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετήσουν την πραγματική οικονομία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και θεωρώ πως η συζήτηση αρχίζει να ξέχναει αυτό το πράγμα, καθώς έχουμε όλο και εντονότερο lobbying ε, των ενδιαφερομένων, γιατί βεβαίως δεν θέλουν να έχουν τόσο ισχυρές απαιτήσει γιατί πέφτει η κερδοφορία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην πέσουμε στην ίδια παγίδα. Και σε σχέση με αυτή την πρόταση θα ήθελα να φέρω κάποια σημεία σημαντικά για μας. Χρειαζόμαστε αρχές διάσωσης οι οποίες θα έχουν ε, μεγάλη διακριτική ευχαίρεια και κάποιες προτάσεις μειώνουν, αν φοβάμαι, τις αρμοδιότητες ε, του συστημικού συμβουλίου, του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Τέλος, πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς για την ιεραρχία των πιστωτών ε, και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Τέτοιον δεν πρέπει να επιτρέψουμε νέες δικαιολογίες για κάποιες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες. Δεν χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ε, των ε, κέντρων offshore από ε, το παράθυρο. Όλα τα μέσα θα πρέπει να υπάγονται σε bail-in χωρίς εξαιρέσεις. Αλλιώς πραγματικά μεταχειριζόμαστε χειρότερα τα δικά μας ε, χρηματοπιστωτικό κέντρα και έχουμε δει στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει bail-in σε μέσα που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες. Και επειδή σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο χρόνος, κατάφερε η Κομισιόν να επιμείνει σε πλήρες bail-in, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Κομισιόν εδώ πέρα άνοιξε την πόρτα για ειδική μεταχείριση τρίτων χωρών. Ε, αυτό πάει ενάντια στην λογική των όσων προτείναμε μέχρι στιγμής. Αυτές οι πρώτες παρατηρήσεις από εμάς και σας ευχαριστώ και αναμένω την καλή συνεργασία στο μέλλον. Και όπως πάντα βεβαίως ε, αυτό το θέμα θα το παρακολουθήσει ο Ερνέστο Ουρτασούν, ο σήμερα απουσιάζει. Thank you. Ε, ευχαριστώ. Είστε έτοιμος κύριε Καμάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ζητώ συγγνώμη που άργησα ή εσείς ξεκινήσατε πιο νωρίς, δεν ξέρω τι από τα δύο συνέβη. Κατά πρώτον να πω και πολύ θα το ξέρετε ότι πολύ συχνά οι συζητήσει αυτές για την διάσωση των τραπεζών και την κρίση τους κοιτάζοντας προς τα πίσω μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Εγώ προσωπικά δεν είμαι βέβαιο στον κάποιοι λένε ότι πρέπει να έχουμε υψηλότερε κεφαλαιοκέ υποχρεώσει και απαιτήσει για τι τράπεζε. Έτσι καλώ τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Κάθε φορά που υπάρχει χρηματοπιστωτική οικονομική κρίση, τα διδάγματα τη κρίση είναι σημαντικά, αλλά η συλλογική μνήμη σιγά σιγά εξασθενεί. Και ο κόσμο λέει δεν θα ξαναγίνουν αυτά, τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα και ξαναγίνονται. Και το δεύτερο που πρέπει να ρωτήσουμε του εαυτού μα είναι τι θα γίνει αν μια τράπεζα πτωχεύσει αύριο. Πώς θα διασωθεί με ε, ίδια μέσα, με άλλα μέσα, χωρίς φορολογούμενο να χρειαστεί να την καλύψουνε. Εάν σκεφτείτε την κρίση του 2007-2008 και τόσα χρόνια μετά την κρίση, 10 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό. Θεωρούμε ότι έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ω προ τι λεπτομέρειε εδώ θα τα, δούμε, θα τη σειρά για τα εργαλεία διάσωσης. Η πρόταση της Επιτροπής να ε, διευθετηθεί η υπαγωγή, η, υπόταξη, με το κρατικό χρέος των κρατών μελών να λαμβάνεται υπόψη, είναι σημαντικό ανάλογα με τα εργαλεία που έχουμε με για τις κεφαλικές υποχρεώσεις. Όμως θα θέλα να το συζητήσω και στην ομάδα μου πριν ε, αποφανθώ περί των λεπτομεριών. πρέπει να δούμε τα τραπεζικά μοντέλα και τα, μοντέλα χρηματοδότηση που λαμβάνονται εδώ υπόψη για να καθοριστούν συγκεκριμένε κεφαλαιοκέ υποχρεώσει. Ω προς το χρονοδιάγραμμα της εξέταση του θέματος είμαι αρκετά διαλεκτικός, αν και πολλοί θέλουν την ταχεία διαδικασία από ό,τι άκουσα. Για τα TILAG και τις ελάχιστε απαιτήσει, τι κεφαλαιοκέ απαιτήσει και για τα στοιχεία και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις, ε, όντω, εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα κριτήρια ιδίω για την ε, επιλεξιμότητα. Τα ήδη υπάρχοντα κριτήρια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά όχι μόνο βάσει των υποχρεώσεων τη επιτροπή, βάσει και των ε, καταστατικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η νομοθεσία είναι αναλογική. Όταν λέω αναλογική, δεν ε, σημαίνει ότι οι τράπεζε θα πρέπει να την ε, σκαπουλάρουν ε, με είδου συμπεριφορών που είχαν και στο παρελθόν. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχέ μπορούν να ζητήσουν υψηλά επίπεδα MRL ελάχιστον δηλαδή απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τι επιλέξιμε υποχρεώσει από τι τράπεζε, αλλά ε, να ξέρουμε και τι επιβάλλουμε στι τράπεζε ανάλογα με το μέγεθό του. Και σε κάθε περίπτωση τι επιμέρου λεπτομέρειε θα ήθελα να τι συζητήσω πρώτα στο επίπεδο τη ομάδα μου. Ω προ την δυνατότητα ανακεφαλαιοποίηση ε, των ε, ε, θεσμών των τραπεζών και την δυνατότητα απορρόφηση των ζημιών, θα πρέπει να κοιτάξουμε εδώ τη μείωση του κόστου και την ενίσχυση τη οικονομική σταθερότητα καθώ και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για του φορολογουμένου. Αυτό θα πρέπει να είναι πάντοτε η βασική μα πηξίδα. Ε, Όμω, επειδή αυτό ισχύει και για τις τράπεζες που την έγινε της Κεντρικής Τράπεζας ε, και για τις υπόλοιπες, θα ήθελα να το δω προηγουμένως με τα μέλη της ομάδας μου, που σίγουρα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά από ότι το δικό μου κράτος μέλος. Ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να συμφωνήσω με την κατεύθυνση που υπέδειξε προηγουμένω ο Φάμπιο Μάζη προηγουμένω για την ανάγκη μια θεωρητικής μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματο ούτω ή άλλω. Διότι αν υπάρχουν τραπεζικέ κρίσει που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ε, με, τα δύο, με το κάθε πόδι σε διαφορετική βάρκα, ε, θα πρέπει εδώ να δούμε τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο, τι θα γίνει σε 60 χρόνια ή αν ακόμα βασιζόμαστε στο μοντέλο Glastinger, ε, που είναι παλιό. Πρέπει να δούμε μήπως αυτό το μοντέλο ακριβώς είναι η αιτία των τραπεζικών κρίσεων, μήπως ε, στην οικονομία σήμερα και στα χρηματοπιστωτικά έχουν αλλάξει κάπως οι συνθήκες και οι απαιτήσει τη πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο και μετά, υπό αυτό το φω, πρέπει να δούμε τα πακέτα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διεθνή πρότυπα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η βούληση, διότι το λόμπι των οικονομικών και των χρηματοποστοτικών υπηρεσιών επηρεάζει πάρα πολύ και την κατάρτιση τη νομοθεσία. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια πρέπει να αναλύσουμε τι διατάξει που έχουμε μπροστά μα, τα στοιχεία του πακέτου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του των εκθέσεων της επιτροπή μας. Οι δύο βασικέ επικριτικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα επικεντρωνόμαστε στην δράση πίστοση, δανειοδότηση δηλαδή, σε σχέση με την οικονομική. Είναι σημαντικά και αυτά. Όμω πρέπει να καταλάβουμε πω κάποια τραπεζικά συστήματα, κάποια οικονομικά συστήματα διαφέρουν από άλλα. Το να έχουμε έναν και μόνο κανόνα που ορίζει ότι κάποιο είναι υγιής αν είναι 1,90 με γαλανά μάτια και 60 κιλά και ζυγίζει 60 κιλά, ενώ κάποιος άλλος που είναι 1,60 είναι 50 κιλά και θεωρείται ότι δεν, δεν εμπίπτει στο σωστό μοντέλο, αλλά παρόλα αυτά είναι υγιής, κάτι δεν πάει καλά. Ε, έτσι πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα κράτη του Νότου, λόγου χάρη όπως στην Ιταλία. Δεν είναι όλα τα πρότυπα ακριβώς ε, ίδια για όλους. Οι τράπεζες δεν μπορούν να πάρουν πιστώσεις, μάλλον να δώσουν πιστώσεις σε κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων και κάποια τραπεζικά μοντέλα τιμωρούνται. Τιμωρούνται για τις οικονομικές τους δραστηριότητες, ενώ είναι διαφορετικό το μοντέλο στην ουσία. Δημιουργείται λοιπόν μια τεράστια στρέβλωση, εάν αφιψηλού από καθέδρας ορίζουμε έναν κανόνα που δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα για δημιουργεί στρεβλώσει και ανισορροπίε. Εδώ λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα αξιολογεί ε, καταλήλω τι ανάγκε ρύθμιση διαφορετικών συστημάτων στην ουσία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώ σφάλουμε. Η πρόταση να προβλεφθούν κυρώσει για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και σε κρατικό επίπεδο, αυτή είναι μια ε, προπόθεση που δεν θα δεχτούμε ουδέποτε με τίποτα. όλοι νομίζω οι εκπρόσωποι κρατών ε, τη Νότια Ευρώπη, διότι θα είχε ένα αντίκτυπο καταστροφικό. Θα κατέστρεφε ε, την έκθεσή μα, ε, την έκθεση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, σε κρατικά ομόλογα, σε κρατικού τίτλου. Είναι μια τεράστια έλλειψη ισορροπία αυτή μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου. Και πραγματικά θα εντείνει και θα οξύνει και άλλο τι εντάσει. με τα πρώτα πακέτα μέτρων ήδη σκεφτείτε σε τι θέση φέρατε τις τράπεζες του Νότου που έχουν πραγματικά τραπεζικά μοντέλα διαφορετικά. Εδώ λοιπόν θα δημιουργηθεί περαιτέρω ένταση και καταστάσεις αντιπαράθεσης. Θα πρέπει λιγάκι λοιπόν να ε, δείξουμε ψυχραιμία και να αξιολογήσουμε σωστά τα διάφορα στοιχεία τη έκθεση, να δούμε ποιε είναι οι σωστέ κατευθύνσει ανάλογα με τα διάφορα τραπεζικά μοντέλα. Έπειτα για τα στοιχεία του BRRD, ε, αυτά που ανέφερε και ο εισηγητή, θα τα δούμε μετά, αλλά σε ό,τι αφορά την ε, ε, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, εάν θέλουμε ένα σύστημα που περνάει από τη λογική οι φορολογούμενοι και από τα πληρώνουν ε, τα σπασμένα της κρίσης, τότε Πώ θα γίνει αυτό όταν οι φορολογούμενοι και οι αποταμιευτέ δεν είναι αυτοί που μπορούν να καταλάβουν και να ελέγξουν τι κάνουν οι τράπεζε. Δεν είναι πολύ σωστή αυτή η διαχείριση και αδίκω βρίσκονται να πληρώνουν τα σπασμένα του. Αυτά που το τραπεζικό σύστημα έκανε μαζί ενδεχομένω με την ε, συνενοχή των πολιτικών και όσων έχουν οργανώσει αυτό το σύστημα. Επιπλέον, η BRRD και η διάσωση με τα ίδια μέσα, τον Μπεϊλίν δηλαδή, είναι πολύ συχνά σε αντίφαση με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα προστασία. Αυτό λοιπόν κατά με δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς όπως προβλέπετε τώρα, αλλά τελείως να εξαλειφθεί. Διότι όπως είδαμε και στο παρελθόν δεν μπόρεσε να αποτρέψει καμία οικονομική κρίση. Κατά την Δική μας λοιπόν αξιολόγηση, αυτές είναι οι βασικές επικρίσεις. Έπειτα πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να προχωρήσουμε στη συζήτηση και να μπορέσουμε και εμείς να υποβάλουμε τις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ. Ακούστε. Ήμασταν ε, στο σκέλος BRRD. Αλλά οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούσαν το δεύτερο σκέλος. Έτσι, το λέω απλά για να γραφεί στα πρακτικά. Τον κύριο δεν τον βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Άρα, η Ντανούτα Χούπνερ στο ΚΑΤΣΔΙ. the Eye. Ευχαριστώ. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να κάνω μια ερώτηση που μάλλον πρέπει να απευθυνθεί προς την Κομισιόν και σχετίζεται με το ότι πέρσι τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έκανε μία σύσταση για να αλλάξει η βάση για το επίπεδο στόχου των ε, εθνικών ε, συστημάτων διάσωσης ε, για να καλύπτουν όχι μόνο τις καταθέσεις αλλά όλα τα ανοίγματα των τραπεζών. Αλλά η Κομισιόν δεν το υιοθέτησε αυτό στην τροπολογία του BRD και έχουν εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είχε μερικά πολύ πιστικά επιχειρήματα για να γίνει κάτι τέτοιο και το ερώτημά μου προς την Κομισιόν είναι να ασχοληθούμε, να μας απασχολήσει ή έχει ξεκάθαρα επιχειρήματα η Κομισιόν και καλό είναι να μην ε, ασχοληθούν οι εισηγητές. Ευχαριστώ. Ασηγητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια. Κοιτάξτε, για την ιεράρχηση και τις απαιτήσει της, αν τα κάνουμε λάθος, δεν θα επιτύχουμε αυτό το οποίο θέλαμε με το BRD, ότι όλο το χρέος υπόκειται σε Μπέιλιν. Και θα αντιστρέψουμε αυτό το οποίο είχαμε επιτύχει με την σχετική οδηγία. Και θα ήθελα να επισημάνω κάτι το ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στην εφαρμογή της οδηγίας αυτής είναι, όπως το είδαμε στην πραγματική ζωή, είναι το ότι όταν δεν είχαμε ενημέρωση από τους πολίτες και τους καταθέτες ότι τα λεφτά τους ήταν εκτεθειμένα σε αυτόν τον κίνδυνο. Και έως αν δούμε την συζήτηση για μια Ιταλική τράπεζα. Αυτό ισχύει και νομίζω πως είναι σημαντικό ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας ε, δισταγμός πως όλο το χρέος στην τράπεζα υπόκειται σε Μπέιλιν. Και εδώ πέρα συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο Σβεν Όμως το θέμα ε, της τρίτης χώρας ίσως είναι πιο περίπλοκο λόγω ε, νομικών ζητημάτων. αλλά η αφετηρία είναι αυτή. Αυτό το οποίο είπε ο κύριο Περέρα επίσης είναι σημαντικό. Να μπορούν να λειτουργήσουν οι τράπεζες και να χρηματοδοτούν επενδύσεις. Και πρέπει να πω ότι Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ισχυρή οικονομία και ισχυρών τραπεζών. Γιατί βλέπουμε σε όλε τι κρίσει ότι μια αφετηρία για τι κρίσει στον τραπεζικό τομέα είναι η ασθενή οικονομία. Ε, όχι ο μόνο λόγο. Τι, εντάξει, μπορεί κάποιες τράπεζες ε, να έχουν κακοδιαχείριση ή να έχουν αναλάβει υπερβολικούς κινδύνους. Αλλά σε γενικέ γραμμέ ε, πρέπει να έχουμε ισχυρέ τράπεζες για μια ισχυρή οικονομία, αλλά και ισχυρή οικονομία και να έχουμε ισχυρέ τράπεζες Είναι αλληλένδετα. Ε, πρέπει να επιμείνουμε. Ο Καμάλ ανέφερε ε, το θέμα του ότι λέμε αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι κάθε φορά είναι διαφορετική και είναι νομίζω, αλλά ε, Βεβαίω ε, συμφωνώ και με αυτό το οποίο είπατε, ότι, δηλαδή, γιατί θα υπάρξουν νέες τραπεζικές κρίσεις. Κάποιοι λένε ότι κάθε δέκα χρόνια θα γίνεται αυτή η δουλειά, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να έχουμε και αυτό δεν είναι θέμα το εάν θεωρούμε ότι η νομοθεσία ε, είναι υπερβολική ή όχι. Εγώ θέλω να υπάρχει ενημέρωση στην τράπεζα, στους, στην αγορά, με συγχωρείτε, στους επενδυτές, σε όσους εμπλέκονται στην τραπεζική αγορά, ότι το χρέος ε, μπορεί να υποστεί bail να υπάρχει μια ξεκάθαρη ιεραρχία επίσης και δεν θέλω αυτή η ιεραρχία να αποφασιστεί κατά τρόπον ώστε κάποιος να θεωρεί ότι δεν θα υποστει η Μπέιλιν. Αλλά χρειάζεται μια αυστηρή ιεραρχία και είναι σημαντικό κομμάτι του BRD γιατί δημιουργώντας έτσι αυτή την ενημέρωση ε, δημιουργούμε σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα και μετά χρειαζόμαστε σταθερούς κανόνες για να αντιμετωπίσουμε το θέμα γρήγορα. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκουλάρ. και να πω και κάτι άλλο. Μπορούμε να πούμε ότι η οδηγία BNRD ε, λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Αλλά ε, είναι δύσκολο βεβαίω να πούμε κάτι τέτοιο, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την οδηγία στην εφαρμογή και τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα είναι κατά κάποιον τρόπο το η ενημέρωση θα έλεγε κανεί για το μέλλον ότι οι επενδυτές θα ξέρουν ότι όταν επενδύουν σε μια τράπεζα βεβαίω τα λεφτά τους ε, διατρέχουν κινδύνους. Σα ευχαριστώ λοιπόν και για τη συνεργασία με την υπόλοιπη διαπραγματευτική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εσύ ήταν. Και βεβαίως πράγματι υπάρχει διαφορά bail-in μεταξύ διάσωσης ε, τράπεζας ε, και μιας προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης. Και τώρα περνάμε, ναι. Θα έδινα τον λόγο στην Κομισιόν στο τέλος ε, και των δύο συζητήσεων. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να περάσω στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο πακέτο και τον εισηγητή τον Πέτερ Σίμον. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για το ότι σήμερα έχουμε αυτά τα δύο θέματα ταυτόχρονα γιατί όπως είπε ο πρόεδρος είναι ε, το λογικό αυτό να δούμε παράλληλα και σε μία θα έλεγα κοινή συζήτηση τα θέματα αυτά πριν ε, υποβληθούν τα σχέδια των εκθέσεων. Το καλύτερο θα ήταν, το χειρότερο με συγχωρείτε, θα ήταν να μην ε, ε, έχουν συντονιστεί οι δύο εκθέσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε τις συζητήσεις και το πώς συνδέονται αυτά τα ζητήματα. Στην μεταρρύθμιση της Οδηγίας και Φυλακών Απαιτήσεων 4 και της CRR ε, δεν είναι μόνο λόγω του μεγέθους και της τεχνικής φύσεως, αλλά και λόγω της σημασίας της για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Μιλάμε για κάτι το οποίο πραγματικά μας απασχολεί εντατικά και επίκαιρον, γιατί υπάρχουν πολλές καινοτομίες που αποφασίστηκαν στις ε, επιτροπές της Βασιλείας, αλλά αν είχαμε κατευθυνθεί σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και υψηλότερη ποιότητα κεφαλαίου ως αντίδραση στην ε, οικονομική κρίση, τώρα δίνουμε το βάρος στην οδηγία κεφαλαϊκών απαιτήσεων 5 θα έλεγα ή στην CRD2 στον επανυπολογισμό και στην υποχρεωτική εφαρμογή διαφόρων διατάξεων ε, και του λόγου μόχλευσης και βεβαίως της αρχής της αναλογικότητας. Επιπλέον θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ενώ όλες οι τραπεζικές αγορές στα κράτη-μέλη επηρεάζονται και βεβαίως σχετίζονται και με την κατάσταση σε όλα τα κρατη Εγώ έχω αυτή τη στιγμή συζητήσεις με εκπροσώπους πέντε διαφορετικών χωρών και ο κάθε ένας έχει ένα διαφορετικό σημείο στο οποίο θέλει να δώσει έμφαση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε στο ευρύτατο αυτό το θέμα να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη στο μέτρο του δυνατού. Πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό έχει σημασία ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων, να κάνουμε κάτι το οποίο θα ε, έχει ένα μεγάλο βαθμό συμφωνίας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε Ποιε πιθανότητε επιτυχία στον τριμερή διάλογο. Λοιπόν, να περάσω τώρα στα συγκεκριμένα θέματα. Αναλογικότητα. Θεωρώ πως είναι γενικά γνωστό ότι ειδικά οι μικρότερες τράπεζες ε, υποφέρουν, θα έλεγα, περισσότερο από το ρυθμιστικό πλαίσιο από ότι οι μεγαλύτερε. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχα πριν από λίγε εβδομάδε όπου είχα απέναντί μου εκπροσώπου των τραπεζών και μου είπαν ότι ε, η τράπεζά μας έχει 56 άτομα προσωπικό και έχουμε δύο άτομα που ασχολούνται μόνο με, τα διοικητικά. Και με αυτά που μας κάνετε θα αναγκαστούμε να συγχωνευτούμε με μια άλλη τράπεζα όχι για λόγους οικονομικούς αλλά γιατί δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε ε, όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο ως μικρή τράπεζα. Για μένα λοιπόν ενδιαφέρον είναι ε, και αυτό μου το είπαν από πολλές χώρες ε, ότι υπήρχε κριτική για το διοικητικό αυτό ε, βάρος το οποίο αντιμετωπίζουν καλύτερα οι μεγάλες τράπεζες γιατί έχουν σχεδόν τα ίδια δεδομένα αλλά με διαφορετική σύνθεση ε, και σε διαφορετικό χρονικό σημείο που τους ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ΕΜΠΑ, η Μπάφιν στη Γερμανία ή όπως λέγεται η οπως λεγεται αρχή και ε, μας είπαν πως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο για να υπάρξει κάποιος συντονισμός για να μην στέλνουν δύο και τρεις φορές τα ίδια πράγματα, κάτι το οποίο απασχολεί πολλούς πόρους και προσωπικό. Ε, λοιπόν, όταν μιλάμε για αναλογικότητα, για μικρότερες τράπεζες, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε ένα χειρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά ένα πλαίσιο το οποίο θα ταιριάζει στην κάθε τράπεζα, στον κίνδυνο και στις απαιτήσει της κάθε τράπεζας. Αν δούμε την πρόταση της Κομισιόν, έχουμε παραδείγματος χάρη διαφορετικές συχνότητες ε, αναφορών και βλέπουμε μετά το εάν επαρκεί αυτό ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη μέθοδο. Επίσης πρέπει να συζητήσουμε τα κατόφλια που έχουμε ορίσει τώρα για την αναλογικότητα. Πρέπει αφενός να διασφαλίσουμε ότι οι μικρές τράπεζες βεβαίως θα έχουν λιγότερο βάρος, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε παραδείγματο χάρη οι τράπεζες που έχουν μικρούς ισολογισμούς αλλά έχουν μια συστημική ε, σημασία να μην ε, καταλήξουν ε, να αποτελούν έναν μεγάλο κίνδυνο αν μιλάμε για ένα μικρό κράτος μέλος. Όσον αφορά λοιπόν τα κατόφλια. Θα πρέπει να δούμε πως τα ποσοτικά κριτήρια που περιέχονται στην πρόταση της ε, Κομισιόν ε, πώς θα μπορούσαν να γίνουν ποιοτικά και να είναι εναλλακτικά ή σωρευτικά. Να δούμε δηλαδή αν θα υπάρξει από εκεί κάποια διευκόλυνση ή όχι. Κατόπιν θα ήθελα να αναφερθώ στο NSFR, το Net Stable Funding Ratio. Το πλαίσιο κάλυψης ρευστότητας έχει ήδη εφαρμοστεί όπως είπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο σημαίνει ότι θα εισαχθεί ένα υποχρεωτικό νούμερο το οποίο θα αφορά την σταθερότητα και σημαίνει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα αναχρηματοδότησης για ένα έτος. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις προσπάθειες της Κομισιόν να συνδέσει τα στανταρτής Βασιλείας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εδώ πέρα έχουμε ακριβώς την προτιμήση των σταθερών καταθέσεων, των ρέπος και βεβαίως της υψηλής ρευστότητας. Και εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε μήπως οι προσαρμογές αυτές στο σύνολό τους είναι σωστές, μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επιπρόσθετες ρυθμίσεις ε, για να δούμε τις οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια πάρα πολύ καλή αφετηρία με την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά τον λόγο μόχλευσης. Το επόμενο θέμα η εισαγωγή ενός υποχρεωτικού λόγου χρέωσης ε, μέχρι 3% νομίζω πως είναι πάρα πολύ θετική γιατί η η Κομισιόν έχει, έχει εφαρμόσει και τις προτάσεις της Βασιλείας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες μέσω της εξαίρεσης των περαιτέρω πιστώσεων σε δημόσιους φορείς, ε, επίσης ε, τις πιστώσει μεταξύ των ομίλων και Βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε εδώ τις λεπτομέρειες ε, και τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής αγοράς. Ένα άλλο θέμα είναι οι ε, τράπεζες ε, εκείνες αναπτυξιακές τράπεζες καθ' αυτές που έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Θεωρώ πως οι αναπτυξιακές τράπεζες διαφέρουν από τις κανονικές τράπεζες και θα πρέπει να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση θα έλεγε κανείς αν προκύπτει από τον ισολογισμό τους ότι απλά θα έλεγα κατευθύνουν τα κρατικά κονδύλια είναι δημένοι στον ισολογισμό τους, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν κάποιον κίνδυνο για τις αναπτυξιακές αυτές τράπεζες. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό νομίζω γιατί η ιδιαίτερη σημασία των αναπτυξιακών τραπεζών για την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη μας είναι νομίζω γνωστή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προτελευταίο θέμα. Εδώ και στην παλιά CRR και στην οδηγία Κεφαλαίων απαιτήσεων Τέσσερα νομίζω πως είχαμε αυτή την έκπτωση 23% για τις πιστώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και γράφει τώρα η Κομισιόν πως προσεχώς θα υπάρχει έκπτωση 50% για τις πιστώσεις πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι το θετικό, αλλά πρέπει να συζητήσουμε το εάν επαρκεί σε μια Ευρώπη στην οποία ε, θα πρέπει να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι παραδοσιακά η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη προέρχεται από τον τραπεζικό τομέα και μπορούμε να είμαστε νομίζω λίγο πιο θαραλέοι από την πρότασή της Κομισιόν. Τελευταίο θέμα, κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα των υποδομών Εδώ πέρα μιλάμε για επενδύσεις σε υποδομές ε, που επίσης προβλέπεται ότι θα έχουν μια έκπτωση κινδύνου, ε, κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, αλλά πρέπει να δούμε ε, για ποια έργα μιλάμε σύμφωνα με τον κατάλογο των κριτηρίων Παραδείγματο χάρη, διαβάζοντας, δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα προωθηθούν μόνο τα έργα εκείνα τα οποία είναι αναχρηματοδοτήσιμα. Εκτός αν είναι το σημάδι ότι οι δημόσιες υποδομές δεν είναι αναχρηματοδοτήσιμες. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά τα έργα, πώς ε, χρειάζεται μια ιδιαίτερη έκπτωση. Επίσης, ε, ο θέμα των υποδομών μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε πολιτικά μηνύματα και υπάρχουν στο θέμα αυτό δισεκατομμύρια επενδύσεων που κανείς δεν ξέρει πώς θα χρηματοδοτηθούν όλοι μιλάνε για ακίνησία αλλά κανείς ε, για την ηλεκτρική με συγχωρείτε κινητικότητα αλλά κανείς δεν ε, μας λέει πώς ακριβώς θα μπορέσουν να γεμίσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και να φορτίσουν αν δεν έχει ο καθένας ένα γκαράζ στο σπίτι του που θα βάλει την πρίζα. Ένα απλό θέμα που θα πρέπει νομίζω να δούμε μέσω μιας έκπτωσης για να διευκολύνουμε ακριβώς την πίστοση στον τομέα αυτών. Τέλος, ακόμη πιο τέλος, έχουμε το IFRS 9, τα, τις διεθνείς αυτές προδιαγραφές ε, για το πώς γίνονται οι χρηματοπιστωτικές αναφορές. Λοιπόν, αν ε, προχωρήσουμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, έχουμε θέσει ως στόχο να έχουμε μία έκθεση ε, με την οποία θα έχουμε συζητήσει με όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς ε, στις 8 Ιουνίου, κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε φέτος ακόμα, ελπίζω, αλλά νομίζω ότι σημασία εδώ πέρα έχει η ποιότητα και όχι η ταχύτητα. Θα δούμε λοιπόν το εάν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την ημερομηνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι η ποιότητα προέχει. Αλλά είναι θετικό αυτό που είπατε, ότι εξετάζετε, μάλλον είστε θετικά διακείμενος. Ε, ενδεχόμενα σε, διαδικασία, σε ταχεία διαδικασία, fast track. Θα το δούμε και με βάση τη συζήτηση και θα δούμε πώς προχωράμε και τι θα κάνουμε. Εκ του κύριου Κάρας, ο Μπούρκα Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ε, για προσωπικούς λόγους χρειάστηκε να επιστρέψει στη Βιέννη ο κύριος Σότο και μου ζήτησε να αναγνώσω εγώ τη δική του δήλωση. Είναι ισχυώδηση για τις εκ του ΕΛΚ. Χαιρετίζει αυτό το περιεκτικό πακέτο της 31ης Νοεμβρίου του 2016 της Κομισιόν θέλουμε ε, να έχουμε την Τραπεζική Ένωση, άρα πρέπει να έχουμε ένα εγχειρίδιο κανόνων. Αυτό είναι το θεμέλιο. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά επαναλαμβάνονται, ή μάλλον στο Διεθνές Μουσικατικό Ταμείο αναφέρουν ότι υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι Έχουμε κάποια μηνύματα από τη ΣΥΠΑ, τα δύο διατάγματα του Πρόεδρου Τραμπ. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις του Brexit. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να μας ε, ε, βγάλουν από το δρόμο μας να λύσουμε τα προβλήματα που έδειξε σε αυτή την κρίση. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. του Μαρκάρας σε ό,τι αφορά το CDR και το ε, CCR. Υπάρχουν ακόμη κάποιες επιφυλάξεις και θα πρέπει να ε, θα πρέπει λοιπόν να, φροντίσουμε, ναι μην ξεκίνησε το αυτοκίνητο, να μην σπάσει το λάστιχο στη μέση του δρόμου. υπάρχει αυτή η απέτηση για την ε, ρευστότητα. Πρέπει να βελτιστοποιήσουμε όμως τις διατάξεις. Επίσης, σε αυτούς τους supporting factors, ο κύριος Κάρας εδώ και χρόνια ζητάει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο κάτι τέτοιο. Αυτή η στόχευση, η στάθμιση, με 25% θα διευκολύνει την χρηματοδότηση στην ενέργεια, την καινοτομία, τις μεταφορές, ε, την ε, παιδεία, την έρευνα. Σε ένα άλλο σημείο. Είναι ιδιαίτερο ο Ευρωπαϊκό Τραπεζικός Τομέας και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε διάφορα σημεία, όπω ό,τι αφορά την ευελιξία και σε ό,τι αφορά το δεσμευτικό δίκτυο καθαρή σταθερή χρηματοδότηση. Είναι λογικά αυτά που προτείνει η Κομισιόν, αλλά σε κάποια σημεία δεν πηγαίνει ε, ακριβώς εκεί που θα ήθελα. Δεν πηγαίνει τόσο μακριά όσο θα ήθελε ο κύριος Κάρας η προτάση της Κομισιόν. Σίγουρα χρειαζόμαστε κανόνες για όλες τις τράπεζες. Η πρακτική όμως δείχνει ότι έχουμε αφενός τις ε, ε μικρότερες τράπεζες και αφετέρου τις μεγαλύτερες, οι οποίες είναι πιο αποφασιστική σημασία. Άρα πρέπει να υπάρχουν, ε, να λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος. Υπάρχουν γυναικές επιχειρήσεις, ε, μικρές τράπεζες έχουν ε, διαφορετικό προφίλ κινδύνου και διαφορετικές ε, διαπλοκές. Οι αναπτυξιακές τράπεζες έχουν έναν κοινωνικό ρόλο, διαφορετικό ρόλο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και βέβαια πάντοτε έχουμε και το εξή πρόβλημα. Μιλάμε μεν για αναλογικότητα, αλλά υπάρχουν διαφορετικές εποπτικές αρχές και διαφορετικά αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ένα σωστός ορισμός και από την εποπτική πλευρά και από την ρυθμιστική πλευρά. Θα πρέπει να γίνει προσαρμογή σε ό,τι αφορά την, προσαρμο... την ε, πληροφόρηση. Αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται διάφοροι παράγοντες, όπως είναι η κίνδυνη και η πολυπλοκότητα του εκάστοτε ιδρύματος ε, και σε ό,τι αφορά και τον ισολογισμό και τις Σε ό,τι αφορά το διοικητικό τομέα. Ένα ενοποιημένο σύστημα πληροφόρηση θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό. Στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τον Νότο Μαρκάρα, το θέμα είναι να βρεθεί σωστή ισορροπία για την αποτελεσματική εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων και κανόνων πρέπει να υπάρξει η σωστή αναλογικότητα για τα μικρότερα ιδρύματα, τις μικρότερες τράπεζες, σε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, κεφαλαϊκή επάρκεια και επίσης ευρωπαϊκή εναρμόνιση, έχουμε το TILAC, έχουμε το MRL και αυτά θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και αν χρειαστεί κάποιοι εκτακτοί κανόνες. Και στόχος είναι βέβαια να μειωθεί ε, ή να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός. Στόχος ε, είναι η ασφάλεια δικαίου. Έχουμε λοιπόν ένα μαραθώνιο ε, στο πλαίσιο της Ιερακής Βασιλείας και θα συνεργαστεί ο Τμακάρας και με τον Πέτερ Σίμων και με τους σκιώδεις mm. εισηγητές. Thank Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για την ομάδα ECR, ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεργαστώ και εγώ με τον κύριο Σίμων και τους άλλους και όλους Η ομάδα μου συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις και καλωσορίζει την ε, μεταφορά των ε, διεθνών προτύπων στο CRR2 και στο CDR5. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, ε, δεν θα είχαμε πρόβλημα, όμως η Κομισιόν βλέπω ότι παρεκκλίνει από τις αρχές της Βασιλείας σε ό,τι αφορά το fast track, γιατί τη μεταβατική περίοδο. Ήδη είμαστε πριν από τον ε, Ιανουάριο του 2018, αλλά αυτό αν το ακολουθήσουμε θα επηρεάσει τις αγορές. Καλό είναι λοιπόν τα πρότυπα διεθνής ε, χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης να ε, διαιρεθούν, να βγουν από, τις, ε, από τη δέσμη αυτή. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο 1 για να μην έχουμε καθυστερήσει και σύγχυση. Και ελπίζω και ο εισηγητής να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Καλό είναι αυτό ο δείκτη καθαρή σταθερή χρηματοδότηση, αλλά η απόφαση τη Κομισιόν με ανησυχεί για τα κρατικά ομόλογα. Ε, Του βάζει μηδενική στάθμιση κινδύνου. Το πρωί αμφισβήτησα το θέμα μπροστά στον Επίτροπο Ντορμπρόφσκη. Αλλά δεν απάντησε ουσιαστικά στην ερώτησή μου. Άκουσα αερολογίες αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο. Δεν μου εξήγησε γιατί η Κομισιόν παρεκκλίνει από την απέτηση Βασιλείας για 5%. Μόνο είπα ότι δεν είναι σκόπιμο πολιτικής πλευράς. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει και ένα χρονοδιάγραμμα για να δούμε πώς θα αρχίσουμε να υπολογίζουμε τους αποτελεσματικούς ε, παράγοντες στάθμισης κινδύνων. Και θέλω και μία σωστή αιτιολόγηση. Να ακούσουμε γιατί η Κομισιόν αλλάζει αυτό από το 5% στο 0% για το CRR. Μας, ανησυχεί. Μας ανησυχούν οι απαιτήσει της Κομισιόν για τις εταιρείες. Το 65% μόνο των προτύπων για τους κίνδυνους αγοράς να εφαρμόσουν εταιρείες και αυτό τρεις ε, χρονιές μετά την έναρξη ισχύω. Μα η αξιολόγηση όλη αυτή είχε στόχο να εντοπίσει τις αδυναμίες της νομοθεσίας. Τώρα τον εφαρμόσει τα θεία της δεν σημαίνει ότι λύνεται και το πρόβλημα. Δέχομαι την ανάγκη για τη μεταβατική περίοδο όμως τελικά στο τέλος αυτής της περίοδου θα πρέπει οι υποχρεώσεις να είναι ξεκάθαρες και ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμόζεται 100% το νομοθέτημα. Αν όμως η Κομισιόν δίνει στον εαυτό της ε, την ε, εξουσία να επιμηκύνει την προθεσμία, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Σε ό,τι αφορά το σε 5 με ανησυχούν οι προτάσει Κομισιόν για ενδιάμεσε εταιρείας χαρτοφυλακίου. Δεν έχει γίνει μελέτη αντικτύπου. θα χρειαστεί μεγάλη αναδιάθρωση μεγάλων εταιριών. Και ίσως υπάρχουν και νομικές επιπλοκές και ασυμβατότητες με άλλες χώρες, με άλλες δικαιοδοσίες. Τέλος. Η απέτηση για αυτή τη δημιουργία τέτοιων εταιριών θα αυξήσει το κόστος ε, το επιχειρηματικό των συναλλαγών στην Ευρώπη. Θα μειώσει την ανάπτυξη, θα χαθούν θέσεις εργασίας και δεν θα είναι ελκυστικός ε, τόπος ε, για τους επιχειρηματίες η Ευρώπη. Δεν θα είναι όλα αυτά υπέρ της εξηγένσης όπως νομίζει και λέει η Κομισιόν. Δεν θα, μπορούν να υπάρξει, δεν θα μπορεί να υπάρξει εξηγένση από τις τράπεζες, αλλά θα δημιουργηθούν εντάσεις και μεταξύ των εποπτών. Είπα και στην αρχή ότι η ομάδα μου επικροτεί τις περισσότερες από τις προτάσεις παρόλα αυτά και θα συνεργαστούμε, όπως είπα και παραλαμβάνω, με τον εισηγητή και τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Μας είπατε και για το IFRS, για τα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. κύριος Βάλι, βέβαια, ε, άσκησε κριτική σε ένα μέτρο που δεν υπάρχει. Αλλαγή για τα κρατικά ομόλογα. Εσείς λέτε ότι διαφωνείτε με κάτι, που όμως δεν υπάρχει στην νομοθεσία. Τέλο πάντων, θα το ξεκαθαρίσουμε, φαντάζομαι αυτό, στην πορεία, όταν ακούσουμε την Κομισιόν. Όταν ρωτήσατε τον αντιπρόεδρο τον πρόσφυγε, δεν ήμουν πάρον εγώ προσωπικά. Μακα... Α, η κόρα Βαν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάπω ανησύχησα ότι ξαφνικά έγινα κύριο, αλλά ευτυχώ δεν είναι έτσι. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον κύριο Ζήμων και του υπόλοιπου ε, σκιώδη σε αυτό το πολύ σημαντικό πακέτο. Όλα όσα κάνουμε εδώ σκοπό έχουν να επιτύχουν το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ διευκόλυνση τη πραγματική οικονομία, να δημιουργήσει θέσει απασχόληση και την παραγωγή ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη και από την άλλη την προστασία των καταναλωτών και την αποφυγή συστημικών κινδύνων. Με αυτό το δεδομένο είναι ακόμη πιο σημαντικό αυτό το πακέτο από ότι ε, άλλα, ειδικά ω προς αυτή την παράμετρο. Ο χρηματοπιστωτικό. Ε, είναι διεθνή, έχουμε πιέσει από διεθνή ανταγωνισμό και πρέπει να δούμε το πακέτο αυτό έχοντας υπόψη το δεδομένο που μόλις ανέφερα. Με ε, μια ε, σαφή προσπάθεια να πετύχουμε ίσως κανόνε παιχνιδιού στο διεθνές επίπεδο. Στο βαθμό του εφικτού θα ήθελα η Γενική Αρχή, ίδια υπηρεσία, ίδιος κίνδυνος, ίδιοι κανόνες, να εφαρμόζεται στον βαθμό που μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Ζήμων και ο κύριος Πάλτς αλλά και ο Γκούναρ Χόκμαρκ ανέφεραν ε, σωστά το στοιχείο της αναλογικότητας. Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες μελέτες αντικτύπου όχι μόνο για να αξιολογήσουμε αυτό το πακέτο αλλά όπως είπε και ο Άσλι για να συνδυαστεί με το IFRS 9, ε, το IFRS 9, τα διεθνή πρότυπα δηλαδή, και την Βασιλεία. Και να βλέπουμε ξεχωριστά με το κάθε νομοθέτημα, αλλά και το συνδυασμό τους. Χρειάζεται μια ε, συνολική μελέτη αντικτύπου για συγκεκριμένα τμήματα συγκεκριμένων κλάδων, συγκεκριμένων περιοχών. Όταν συζητήσαμε ε, για τους κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας είδαμε τι διαφορές υπάρχουν τότε. Με μια γενική μελέτη αντικτύπου ε, δεν βγάζουμε νόημα, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, όταν έχεις τα πόδια σου στο φούρνο και το κεφάλι στο ψυγείο, έχεις ε, καλή μέση θερμοκρασία, αλλά δεν πάνε όλα καλά και στις δύο πλευρές. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς αυτά λειτουργούν στους διαφορετικούς τομείς ταυτόχρονα. Μια άλλη γενική παρατήρηση είναι ότι εφόσον ε, έχουμε πίεση από το διεθνή ανταγωνισμό, η ψηφιοποίηση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι πανταχού παρούσα. Αργότερα θα συζητήσουμε και την, την έκθεση ΦΙΝΤΕΚ την έκθεση FinTech συγκεκριμένα, και να δούμε, ε, το να δούμε κατά πόσο αυτά τα νέα μέτρα θα είναι φιλικά προς την καινοτομία. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο κλάδο θα πρέπει να κάνει τεράστιε επενδύσει για να παραμείνει ανταγωνιστικό σε αυτόν τον ψηφιοποιημένο κόσμο και την κοινωνία. Επί των ε, λοιπόν λεπτομεριών, ε, ευχαρίστω να τη συζητήσω μαζί σα και στο μέλλον, αλλά γενικέ μου παρατηρήσει για την αρχή τη συζήτηση ήταν αυτέ ακριβώ. Σα ευχαριστούμε και τώρα ο Ματ Κάρθη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και την, της πρόταση, την πρόταση της Κομισιόν καθώς ήταν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση αλλά νομίζω πως υπάρχουν τομείς όπου δεν πηγαίνει αρκετά μακριά στα υφιστάμενα προβλήματα. Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το πρόβλημα των τραπεζών too big to fail από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να διαχωρίσουμε την λιανική τραπεζική από την επενδυτική τραπεζική και θα καταθέσουμε εμεί σχετικές τροπολογίες που επίσης θα ζητούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις άλλη ανησυχία που έχουμε αφορά ακριβώς αυτό τον λόγο μόχλευσης μόνο 3%. Θεωρούμε πως ο λόγος μόχλευσης είναι πολύ ε, καλύτερο μέτρο της ε, θέσης που βρίσκεται η κάθε τράπεζα και έτσι θα μπορέσουμε νομίζω να καταλήξουμε σε μια ε, καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού σταθμισμένα ανάλογα με τον κίνδυνο και επίσης είναι πολύ πιο εύκολο να το επιτηρούν οι ρυθμιστικές αρχές. Αλλά πρέπει να είναι πάνω από το 3% ειδικά για τις συστημικά σημαντικές ε, τραπεζές. Π.χ. το 12 πρότεινε ο ένα λόγο μόχλευσης 5% και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε πει πως το 5% θα είναι δύο φορές ε, πιο εποφελέ από το 3% στο να μειωθεί η πιθανότητα χρεοκοπίας μιας τράπεζας. Επίσης, ε, η συνολική ικανότητα απορρόψης ζημιών έχει θεωρηθεί ως ένα μέσο να επιλύσουμε το πρόβλημα των τραπεζών που είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν, αλλά όπως σας είπα δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επίσης η BRD έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο να αποφεύγουμε διασώσεις με τα χρήματα των φορολογουμένων. Και βλέπουμε το τι γίνεται στην Ιταλική τραπεζική κρίση, ειδικά μέσω της προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όποιον θέλει να το δει πως δεν μπορεί να συνεχίσει η διάσωση με λεφτά των φορολογουμένων και υπάρχουν πάρα πολλά παραθύρα και γενικά θα λέγαμε πως ε, πρέπει να αυξηθούν οι κεφαλαϊκές απαιτήσει αντί να εφευρίσκουμε νέες πορύπλοκες έννοιες όπως το τίλακ που υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι δεν θα λειτουργήσουν όταν υπάρξει κρίση. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίω πως δεν υπάρχει πλειοψηφία για να αυξηθεί το κεφάλαιο επίπεδου 1, οπότε θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά τις προτάσεις. Επίσης έχουμε κάποιες ανησυχίες για το ότι το υφιστάμενο επίπεδο TILAC δεν επαρκεί για να μειωθεί ο αντίκτυπος της επόμενης τραπεζικής ε, κρίσης. Αυτή τη στιγμή μόνο 13 ε, τράπεζες με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύπτονται, ενώ οι υπόλοιπες ε, τράπεζες που είναι εξίσου όμως ε, συστημικής σημασίας ε, θα καλύπτονται από το καθεστώς MREL ε, την ελάχιστη απέτηση ιδίων κεφαλαίων και πλέξιμων κεφαλαίων ενώ και άλλες τράπεζες θα μπορούσαν να έχουν εξίσου καταστροφικά αποτελέσματα. Τέλος, για την έκθεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υποδομών θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να βασίζονται στις τράπεζες αυτό είναι δουλειά της μακροοικονομικής πολιτικής και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε μικρο. πολιτική δεν θα λειτουργήσει. Επίσης, ε, ταυτόχρονα βεβαίω θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις απαραίτητες φορολογικές πολιτικές ε, και τότε βεβαίω αυτό θα λειτουργήσει μόνο αν υπάρχουν και κατάλληλες μακροοικονομικές πολιτικές και σταματήσουν οι πολιτικές λιτότητας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες επίσης οδηγούν τις τράπεζες στο να αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους. Ήθελα λοιπόν να υιοθετηθούν αυτές οι προτάσεις μας και νομίζω πως είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Σβέν Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. αφού έχουμε γερμανόφωνη συγκεκριτή θα τα πω γερμανικά και αφού και ο πρόεδρος ε, φαίνεται ότι επιδίδεται στην ε, άσκηση της γερμανικής γλώσσας και αυτός αστείο ήταν τέλο πάντων ουσιαστικά είναι πολύ σοβαρό το θέμα θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτερ Ζήμωνα ε, που έχει κάνει αυτές τις προτάσεις ε, και μπορούμε έτσι να κάνουμε έναν απολογισμό του τι έχουμε πετύχει με την τραπεζική νομοθεσία μετά την κρίση. Και νομίζω ότι είναι ένας ειλικρινής απολογισμός ε, και περιλαμβάνει αυτός διάφορα στοιχεία και θα πρέπει να τα αναλύσουμε και να δούμε και τι αποτελέσματα έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε λοιπόν από τη μια πλευρά ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση σε διάφορα σημεία να χαλαρώσουμε λίγο τα ενία και περιέργως σε οποιαδήποτε συνάντηση έχω και κάνω τα σχετικά ερωτήματα το χρηματοπιστωτικό τομέα, μία ε, κατεύθυνση ε, εξέρουν ότι εξαιρέσεις, ε, κάτι τα κτλ. Επομένως, ε, αυτό το, αυτήν εδώ δεν πρέπει να την ακολουθήσουμε. Στην ανάλυση μας θα πρέπει να δούμε οι κανόνες ε, που δεν έχουν ακόμη πετύχει το στόχο τους και από την άλλη πλευρά που ε, προκαλέσαμε και ζημιά, σε ποιους τομείς ενδεχομένως προκαλέσαμε ζημιά. είναι νομίζω η σαφής εικόνα ότι έχουμε ε, μια νομοθεσία η οποία δεν έχει καταφέρει να είναι η σωστή και χρυσή τομή σε όλες τις περιπτώσεις τελικά το εννοούμε ε, και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Είδαμε τι έγινε στην Ιταλία, είχαμε τη συζήτηση για την Deutsche Bank. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα το στόχο μα και γι' αυτό θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσο και ο δίκη τη μόχλευση, αυτά τα όρια χρέωση είναι υψηλά. Αυτό το 3% είναι αρκετά υψηλό και από την άλλη πλευρά. Όταν μιλά κάποιο με τι πιο μικρέ τράπεζε, ε, πολύ πιστικά λένε αυτό ακριβώ ε, που είπε και ο εισηγητή, ότι δηλαδή διάφοροι δημόσιοι φορείς, εθνικοί, ευρωπαϊκοί, ζητούν λίγο πολύ τα ίδια δεδομένα. Παρότι μπορεί να μην πρόκειται κανένα συστημικά σημαντικό ε, φορέα. Αυτό είναι διαφήμιση ε, και ε, βούτυρο στο ψωμί των αντιευρωπαϊστών. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο είπε και ο Πέτερ Ζήμων ότι μαζί θα πρέπει να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό, το σωστό απολογισμό. Να κάνουμε πιο πολύ για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επίσης, να εξαλείψουμε την στη γραφειοκρατία. Δεν είμαι κατά να μιλήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις για, για πρόσθετες εξαιρέσεις, για παράδειγμα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να βασίζονται όχι ε, σε, πολιτική, σε πολιτικές σκοπιμότητες για την έρευνα του τραπεζών, αλλά σε, στη βάση ε, σωστών αναλύσεων να αντιμετωπίσουμε τη, τους κινδύνους, να δούμε αν γίνεται σωστή στάθμιση κινδύνων, να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Αν είναι πραγματική η κίνδυνη, δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε με την τραπεζική ανάπτυξη, ε, ρύθμιση να έχουμε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη. Για... Αμοιβές, επίσης, ένα θέμα τα μπόνους δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ε, πολύ μεγάλη αμοιβή τελικά ε, σε αυτά τα στελέχη. Αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το μακροπρόθεσμο. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Η Κομισιόν έχει ε, προβεί σε κάποιους περιορισμούς. Αυτές οι τόσο αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσει πληροφόρηση και δημοσιοποίηση μικρέ τράπεζε, τράπεζες, τι μικρέ φορέ. είναι τόσο απαραίτητε, Αλλά σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστική σταθερότητα, οι κανόνε για τι αμοιβέ πάνε πολύ πιο μακριά. Υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει με τις οποίες δεν συμφωνούμε για, τις, ε, για τους αγορές. Υπόθηκαν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο εισηγητή ότι θα πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα. Εγώ ε, θα έλεγα να μην βασιστούμε μόνο σε μια ακρόαση. Έχουμε πάρα πολλούς φορείς που θίγονται αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και άλλους παράγοντες ε, που τους αφορά πάρα πολύ χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να ακούσουμε οικονομικούς παράγοντες ε, και πολλούς άλλους, οι οποίοι θα πρέπει να μας δώσουν ε, την εμπειρία τους. Θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω από μια ακροάσεις, να ακούσουμε θυγόμενους φορεί, φορείς, να ακούσουμε και ενός καταναλωτών και άλλους φορείς που έχουν να πούν πράγματα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ισορροπημένη θέση και προσέγγιση, περισσότερη αναλογικότητα από τη μία πλευρά ε, και εξάλληψη αχρέως των ε, ρυθμίσεων, ε, λιγότερη γραφειοκρατία και βέβαια πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στους στόχους μας, μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να μην υποστούμε και να μην λυγίσουμε στις πιέσεις ενός λόμπι. Ευχαριστώ. Βάλει Sì, rapidamente perché ero già intervenuto prima. Ero già intervenuto prima dando le mie considerazioni su entrambi visto che sono Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδη και για τι δύο εκθέσει, οπότε μπορώ να τα πω ίσω μαζί. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο τα κρατικά ομόλογα, από το κρατικό χρέο. αυτό που ήθελα να πω ήταν οι τροπολογίες στο 507 που συζητείται στην Ιταλία για το CRR. Η μπορεί να προβαίνει σε εξαιρέσει ό,τι αφορά το δίκτυο μόχλευση ε, για τα κρατικά ε, ομόλογα που έχουν ε, μηδενικό συντελεστή στάθμισης και μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό συντελεστή. Αυτό θα είχε καταστροφικό αντίκτυπο για τα κράτη της περιφέρειας. Φυσικά τα κράτη του Νότου μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη, αλλά ζητώ τους συναδέλφους να δουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα κρατικά ομόλογα. Για να μην υπάρξουν οι και κάτι που θα ήταν πάρα πολύ αρνητικό. Ναι, ακούστε λοιπόν, εδώ μιλάμε για μελέτη αντικτύπου, μάλιστα. Δεν θα αλλάξει το όριο έκθεση. Είναι μία μελέτη αντικτύπου. Θα το συζητήσουμε σίγουρα το θέμα, γιατί το άρθρο αυτό σίγουρα θα συζητηθεί πολύ. Catch the eye. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή για την άποψη που εξέφρασε για την πρόταση της ε, Κομισιόν. Μια αρκετά μεγάλη πρόταση. Πολλές σκέψεις εκφράστηκαν από τους συναδέλφους ε, και μπήκαν εις βάθος. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο το οποίο πραγματικά έχει αφήσει με κάποιες απορίες το άρθρο 507 η Κομισιόν προτείνει να της δοθεί μια ευρύτατη έντολη και μιλάμε για τα άρθρα 390 και 400 για ακριβώς την έκθεση των τραπεζών στο δημόσιο χρέος. Και βεβαίως το θέμα της ε, προληπτικής αντιμετώπισης ε, των δημοσίων ε, χρεών υπάρχει ήδη στην Βασιλεία αλλά δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία και το Συμβούλιο αποφάσισε να μην καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα πριν κριθούν τα επόμενα βήματα και άρα δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά πριν καταλήξει κάπου η Επιτροπή της ε, Βασιλείας. Θα μπορούσε λοιπόν εδώ πέρα να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τον Ευρωπαίο καταθέτη τραπεζών και μου φαίνεται πως είναι κάπως πρόωρο να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, ειδικά δεδομένου του γεγονότος ε, πως ε, θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή η κατάσταση περισσότερες δυσκολίες για τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα. Επιπλέον το θέμα αυτό το έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά μας για την ε, Βασιλεία το οποίο βεβαίως αφορά και την ε, αναθεώρηση των οδηγιών CRR και CRD για το παγκόσμιο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να μειώσει και όχι να εντείνει τις διαφορές μεταξύ διαφόρων δικαιοδοσιών. Δεδομένου του ότι α, βεβαίως μιλάμε για χρέος το οποίο έχει εκδοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με κίνδυνο ο οποίος τίνει προς το μηδέν. Όπως ε, σας είπα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να κρυθεί το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο λόγω ακριβώς ε, της ε, λεπτής του φύσης. Σας ευχαριστώ. Οπότε. Να δώσω τώρα τον λόγο. Ναι, να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν. Και τον εκπρόσωπό της. Ναι. Ο κύριος Βίτνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά σημεία ακούστηκαν και θα προσπαθήσω να τα αναφέρω. Σε γενικές ε, γραμμές ε, έχουμε αυτό το οποίο αναφέρατε πολύ από εσάς περαιτέρω μείωση του κινδύνου και μιλάμε για υποχρεώσεις για κινδύνους που δεν έχουμε καλύψει ακόμα αλλά ταυτόχρονα, όπως είπατε, πρέπει να φροντίσουμε οι τράπεζες να μπορούν να εκπληρώσουν τον ρόλο χρηματοδότησης της οικονομίας. Οπότε, λαμβάναμε αυτά τα μέτρα μείωσης του κινδύνου και προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια δυνητικά προβλήματα τουλάχιστον βράχη πρόθεσμα στην χρηματοδότηση της οικονομίας και όταν το είδαμε αυτό και βεβαίως όπως πάντα είναι πολύ δύσκολο να δούμε το τι γίνεται όπως ε, παραδείγματος χάρη στο τι έχουν οι τράπεζες στα βιβλία τους ή με το NSFR προτείναμε κάποιες ε, περίοδους μεταβατικές έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε κάποιες υπερβολές από την άλλη βεβαίως αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας οπότε αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε ως ισορροπία ταυτόχρονα βεβαίως όπως αναφέρατε. Έχουμε πολλά μέτρα που αφορούν απευθείας ε, τη χρηματοπιστωτική οικονομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρήσαμε λοιπόν συνολικά πως είναι ισορροπημένος ο συμβιβασμός και θεωρούμε, όπως είπαμε, ότι είναι ένα πακέτο και ως πακέτο πρέπει να το δούμε. Το TILAC είναι κυρίως στην οδηγία CRR, το υπόλοιπο το MRL, η ελάχιστη απέτηση των ιδίων κεφαλαίων είναι στο CRD. Βεβαίως κάποια μπορούμε να τα προχωρήσουμε πιο γρήγορα και νομίζω ότι θα συμφωνήσαμε ότι η ιεραρχία των πιστωτών είναι μια πρόταση και μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα και βεβαίως αναφέρθηκαν ε, και τα διεθνή πρότυπα χρηματοπιστωτικών αναφορών, τα e ΕΑΕΦΡΕΣ 9, οποία θα τεθούν εν ισχύ το 2018 και αυτό θα έχει αμέσως απαιτήσει ε, αντίκτυπο ε, απαιτήσει, απαιτήσεις και μάλλον δεν θα έχουμε και το κείμενο δημοσιευμένο ε, μέχρι την 1η Πρώτου 2018 οπότε και αυτό νομίζω είναι ένας υποψηφίο για να κινηθούμε κάπως γρήγορα. Τώρα για τα ζητήματα που αναφέρθηκαν, η αναλογικότητα, ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι πιο στοχευμένο, είναι αυτό το οποίο είπατε, νέα αναφορές, ε, δημοσιοποίηση, μοντέλα τα οποία είναι ευκολότερα για uh, trading, για να καλύψουμε παρεκκλήσεις. Σκεφτήκαμε και συγκεκριμένα ε, ένα συγκεκριμένο καθεστώς για τις μικρές ε, τράπεζες, αλλά είναι δύσκολο γιατί το θέμα είναι πώς ακριβώς ε, καθορίζεται κάτι τέτοιο. Μετά έχουμε τις τράπεζες αυτές που είναι πολύ μεγάλες, αλλά με απλό επιχειρηματικό μοντέλο που θα πρέπει να έχουν και αυτές την ίδια μεταχείριση. Μετά ποια θα είναι η εναλλακτική μεταχείριση, να μιλήσουμε για πολύ υψηλό λόγο μόχλευσης και να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα. Μετά λέμε τι κάνουμε με την ρευστότητα, οπότε ε, καταλήξαμε σε αυτά τα στοχευμένα μέτρα για την αναλογικότητα, ε, αλλά βεβαίω για τι αναφορέ στην πληροφόρηση είμαστε ανοιχτοί να δούμε πώ θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Και τα ίδια μα είπαν και οι ενδιαφερόμενοι ότι καμιά φορά πρέπει να πούν τα ίδια πράγματα σε διάφορου φορεί. Μπορούμε ίσω να πάμε ένα βήμα πάρα πέρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό εντό του κανονισμού. Επίση το θέμα του δημοσίου χρέους. Η πρότασή μα εδώ δεν αλλάζει την αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ του χρέους του ενός κράτους μέλους και άλλου κράτους μέλους. Ακόμα εκκρεμεί το ζήτημα, αλλά επί της αρχής υπάρχει μηδενική στάθμιση κινδύνου Νομίζω υπάρχει μια παρεξήγηση, νομίζω, εδώ πέρα. Έχουμε τις γενικές διατάξεις για την εθνική διακριτική ευχαίρεια για τη μεγάλη έκθεση. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, γιατί θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε εδώ πέρα να έχουμε περισσότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αλλά τελικά δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο δεν μπορούσαμε να προτείνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, οπότε αυτό το οποίο έχουμε είναι εκθέσεις, αλλά η EBA βεβαίω ε, μας ε, λέει το, στην, εκθέσεις στην EBA και αναφορές για τις μεγάλες αυτές εκθέσεις. Και ένα από αυτά βεβαίως είναι η έκθεση σε κρατικά ομόλογα, αλλά είναι κάτι το πολύ γενικό. Μετά, το θέμα που αφορούσε το bail-in μέσων που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες αυτό γίνεται δεκτό μόνο όμως υπό τον όρο ότι υπάρχει μια ρήτρα συμβατική bail-in στα μέσα αυτά και είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Διάσωσης, το Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο σε περίπτωση διάσωσης ε, και θα υπάρχει βεβαίως έλεγχος οπότε τέθη ένα ε, ζήτημα νομίζω για το Ταμείο Διάσωσης το οποίο δεν κατάλαβα η πρόταση αυτή δεν αφορά καθόλου το Ταμείο αυτό είναι τελείως εκτός του πεδίου εφαρμογής Ευχαριστώ όμω να το συζητήσουμε ενημερώς το τι εννοούσε αυτό που έκανε την ερώτηση και κάτι ακόμα για τον λόγο μόχλευση. Ε, ε, πράγματι δεν έχει τελειώσει η Επιτροπή της Βασιλείας, αλλά ε, αν είχε καταλήξει κάπου η Επιτροπή της Βασιλείας θα το είχαμε βάλει. Μπορείτε να το κάνετε εσείς βεβαίως, να το νομοθετήσετε ε, καθοδόν για τον υψηλότερο λόγο μόχλευσης. Αυτά και ε, όπου μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να προχωρήσουμε αυτά τα έργα. Ευχαριστώ. Είπατε ότι απαντήσατε στα πλέον σημαντικά, όμως και αυτό που ρώτησα εγώ ήταν πολύ σημαντικό. Σας ρώτησα για αυτή τη σύσταση που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή, Κεντρική, για την, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την αλλαγή του μοντέλου, του εθνικού μοντέλου ανακεφαλοποίησης, συγγνώμη πρέπει να στρέφω προς το μικρόφωνο, που ε, δημοσίευσε τον ε, Οκτώβριο η Τροπεζική Αρχή. Αλλά δεν έλαβε υπόψη την ενδεχόμενη αλλαγή που τώρα συζητάμε. Ε, σωστά το πρότεινε, κατάλαβα εγώ λάθος, τη σύσταση ή η αιτιολόγηση της EBA ήταν ε, διαφορετική. Θα περάσουμε δηλαδή την τωρινή πρόσταση στο σύνολο των ε, παθητικών, των στοιχείων του παθητικού, μπορείτε να το σχολιάσετε. Με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Οι συνάδελφοι μου λένε ότι δεν έχει προβλεφθεί τίποτα. Είναι ένα νέο σημείο θα το ελέγξουμε και θα σας στείλουμε την απάντηση. Μάλιστα, ο εισηγητής. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ αναλυτική αυτή συζήτηση και για τα μεμονωμένα σημεία που σχολιάσατε. Χαίρομαι και Αν κοιτάξω γύρω μου, νομίζω ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με, το, με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και τις λεπτομέρειες θα τις βρούμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Υπάρχουν και κάποια ανοιχτά ερωτήματα βέβαια Μέχρι σήμερα πραγματικά δεν με είχαν απασχολήσει, όπως τα κρατικά ομόλογα για παράδειγμα. Πρέπει να σας πω ότι πέρασα αυτή την τυρκουάζ εβδομάδα ε, και ασχολούμουν με τη μελέτη, αλλά δεν άκουσα τίποτα, ούτε μία λέξη, ούτε μία συλλαβή για τα κρατικά ομόλογα και για το άρθρο 507 που αναφέρατε. Πραγματικά εδώ ε, ε, υπάρχουν συνέπειες άμεσες. Μην μπλέξουμε όμως τα πράγματα και μην κάνουμε μια συζήτηση που θα έχει πόρο της πραγματικότητας. Διότι οι κανόνες αυτοί εδώ δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη στάθμιση των κρατικών ομολόγων. Δεν αναφέρουμε τίποτα για την έκθεση σε τέτοιο είδος ομόλογα. Βέβαια, κατά πόσον είναι θέματα που απασχολούν τώρα αυτά τα κράτη-μέλη, θα δούμε αν μπορούμε να περιλάβουμε κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντως, περιμένω και προσβλέπω σε καλή συνεργασία με όλες και όλους Περιμένω τις δικές σας ε, συνεισφορές και η πόρτα μας παραμένει ανοιχτή, όπως και το ε, γράμματο κυβότιο αν, ε, και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν είναι κατηλημένο η τηλεφωνική μου γραμμή, για να συνεργαστούμε και να έχουμε μια καλή θέση. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις διαπραγματεύσεις τριμερή διάλογο να καταλήξουμε εδώ σε μεγάλη πλειοψηφία ως Κοινοβούλιο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε ήδη μια πρόταση. Τον συγκεκριτή για την παρουσία της εκθεσής του, μιλάω τον Πέτερ ε, Ζήμων, 8 Ιουνίου. Θα έχουμε βέβαια ενδιάμεσα hearing και ίσως και άλλη μια ανταλλαγή απόψε. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Χέκμαρκ, το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Κύριο Χέκμαρκ. Ναι, αυτή είναι η πρόθεση μας. Ίσως να είμαστε και μισό βήμα μπροστά από τον Πέτερ, όπως είπα, για να είναι πιο εύκολο ο συντονισμό, αλλά αυτό θα γίνει σε κοινή συνεννόηση μεταξύ μας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα αυτό. Αν όμω πρέπει να συσχετίσετε τη δουλειά σα, καλό είναι να πάτε παράλληλα και όχι να είστε εσεί μισό ή ένα βήμα μπροστά, για να ακολουθεί ο άλλο από πίσω. Και θα έχουμε και πρόβλημα, κύριο Ζήμων, γιατί μπορεί η δεύτερη να μην θέλει να ακολουθήσει. Ή το ανάποδο, λέει ο πρόεδρος. Εγώ θα πρότεινα να κινήσετε εκ παραλίλου. Να έχετε το ίδιο χρονοδιάγραμμα και θα δούμε και με την ταχεία διαδικασία πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά θα τα συζητήσουμε και στις επόμενες συναντήσεις μας. Αυτή τη λύση προτείνω πάντως. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο τη σημερινή διάταξη και να περάσουμε στο επόμενο. Παρακαλώ. 8 Ιουνίου, τέλος πάντων. Είναι η προθεσμία, αλλά θα δούμε. Πώς θα προχωρήσουμε, γι' αυτό δεν σας λέω τις επόμενες ημερομηνίες για το τι θα γίνει με το τέλος του χρόνου. Ας έχουμε το πρώτο, τον πρώτο στόχο, 8 Ιουνίου. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ και τώρα πού είναι το FinTech. Yes was former point six, uh, fintech influence of the... Fintech. Ε, κυρία Φανίβεν Χόιζεν, κόρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευνηδιάζονται νομίζω οι σκιώδεις εισηγητές μου όλοι ε, από το ρυθμό αυτής της συνεδρίασης διότι είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα αλλά θα ευχαριστήσω τους υπόλοιπους σκιώδεις που δεν είναι εδώ για την συμβολή τους και την πολύ καλή συνεργασία που ήδη είχαμε για το θέμα αυτό. Το FinTech είναι ε, πολύ απλό να λειτουργήσει χάρη στα νέα τεχνολογικά μέσα και η έκθεση αυτή ουσιαστικά στρέφεται προς το μέλλον. Είναι μια έκθεση δικής μας πρωτοβουλίας, διότι ενώ ακόμη αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κρίσης με την ισχύουσα νομοθεσία και συζητήσαμε για το CRD και το CRR, παντού στον κόσμο οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και βλέπουμε οι ρυθμιστές να πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν συμβαίνει αυτό μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Σιγκαπούρη. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, όπου οι παραδοσιακά προηγμένες χώρες ε, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Βλέπουμε ότι η πρόσληψη υπηρεσιών FinTech ε, στην ε, στον υπόλοιπο κόσμο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρική, Λατινική, Αμερική, Μέση Ανατολή, είναι περισσότεροι από ό,τι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη και περισσότερο από ότι, ε, περισσότερο στο Silicon Valley ε, από ό,τι στο, μάλλον, περισσότερο στο Ισραήλ από ό,τι στο Silicon Valley. Υπάρχει λοιπόν ε, παρεμβολή εδώ σε όλες τις υπηρεσίες και των μεταφορών και των υγειονομικών και έχει να κάνει αυτό με την τεχνική ευθεία, το υπολογιστικό νέφος, την ε, ψηφιακή ε, χρηματοδότηση. Μια άλλη καινοτόμα τάση είναι ότι άλλοι τομείς που δεν αναμενόταν ως τώρα έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες φορεί που δεν είχαν μέχρι τότε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά. Δηλαδή μπορεί να είναι ασφαλιστικέ, τραπεζικέ υπηρεσίε, αλλά και νεοφυεί και μεγάλε πολυεθνικέ όπω η Apple, η Google και ούτω καθεξή. Με άλλα λόγια, πρέπει να κοιτάξουμε τον κόσμο με ένα νέο βλέμμα, ανάλογο, διαφορετικό από τις, τους διαχωρισμούς τους γεωγραφικούς, τους μεταξύ κλάδων και υπηρεσιών που προσφέρονται θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε ταυτόχρονα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης FinTech, για τα θέματα δηλαδή αυτά, που θα πρέπει να είναι και διασυνοριακό στη διαδρασή του. Δηλαδή όπως ήδη θα έπρεπε να γίνεται στον τομέα του FinTech και η φύσμα ήδη συνεργάζεται με την DG Connect και την DG Grow. Πράγμα θετικό. Είναι πολύ καλό που ήδη συμβαίνει αυτό. Η έκθεση αυτή σκοπό δεν έχει να προσφέρει τεχνικές λύσεις, αλλά να ορίσει μια σειρά από σαφείς παραμέτρους για τη FinTech στην Ευρώπη. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η αρχή της καινοτομίας. Όλος ο ενδεχόμενος αντίκτυπος της τεχνολογίας πρέπει να αξιολογείται καταλήλως. Μια δεύτερη διάσταση, καθότι είμαι φιλελεύθερη, είμαι πάντοτε υπέρ του ανταγωνισμού, του δίκαιου ανταγωνισμού, που σημαίνει ίσου κανονέ παιχνιδιού. Πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι φερόμαστε σε όλου του φορεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτό για μένα είναι μια αρχή απαράβατη. ίδιε υπηρεσίε, ίδιο κίνδυνο, ίδιοι κανόνε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να του εφαρμόσουμε στο δυνατόν περισσότερο. Επίση, πιστεύω ότι η τεχνολογική ουδετερότητα είναι σημαντική. Λόγω χάρη, επειδή συζητήσαμε με το, για το MIFID ήδη πέρσι το καλοκαίρι, και το τι είδου υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να έχουμε επί χάρτου ή όχι. Θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, ψηφιακή μορφή, είχαμε πει τότε. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ελέγχους ε, πειραματικά. Ε, διότι μόνο δρώντας θα διδαχθούμε. Όχι μόνο για τη FinTech βέβαια, αυτό ισχύει ρυθμιστικά από κάθε άποψη και από τη RegTech. Δηλαδή, εάν δεν πειραματιστούμε με αυτό το επίπεδο, με τα εικονικά νομίσματα, με άλλους τρόπους, δεν θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και δεν θα μπορέσουμε ποτέ πραγματικά να έχουμε εποπτεία. Όπως είπα και προηγουμένως, στην προηγούμενη βέβαια συζήτηση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ψηλά πρότυπα προστασία των καταναλωτών και ότι ε, εξασφαλίζουμε χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτέ είναι οι ε, προποθέσει για τι οποίε μιλάμε. Ε, πολλές πολιτικές συστάσεις της έκθεσης έχουν περιληφθεί, όμως η πρώτη είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διότι η δυνατότητα διασύνδεσης είναι σαν οξυγόνο σήμερα, δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς αυτήν και με το να έχουμε όλο ένα και περισσότερο ψηφιακό χαρακτήρα και να είμαστε και πιο ευάλωτοι ω προ το κρατικό χρέο λόγου χάρη. Αυτό μπορεί να σημαίνει και λειτουργικού κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα και μη παροχή υπηρεσιών. Σκεφτείτε τι θα γίνει με 80 εκατομμύρια δολάρια που μπορεί να καταχραστούν από από ε, μια τράπεζα, ένα δισεκατομμύριο λογαριασμού ε, Google μπορεί να, που μπορεί να χακαριστούν. Και πολλέ φορέ χωρί να μένει ίχνος από όλα αυτά. Να ξεχάσουμε λιγάκι τον παραδοσιακό ληστή τράπεζα που μπαίνει με ένα σκούφο στο κεφάλι και ένα όπλο. Τώρα πια οι hacker θα κάνουν όλα αυτά με έναν τρόπο πολύ άνετο, καθισμένοι σπίτι του Και με τεράστιες επιπτώσεις. Και δεν είναι πια το πρόβλημα τα νομίσματα, αλλά τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι κατά κάποιο τρόπο το νέο νόμισμα. Το νέο νόμισμα που έχει πολύ, σημαντικό, ε, πολύ σημαντική διάσταση για αυτό το φάκελο. Μιλάμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα και πολλές προκλήσεις με την τεχνητή ευθεία που μπορεί να συνδυάζεται με την εκμάθηση των μηχανικών μέσων και το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε στοιχεία του παθητικού. Ε, το τελευταίο που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με τις δεξιότητες. Η καινοτομία βασίζεται στο λογισμικό και την τεχνητή ευθεία, της νέες τεχνολογίες, οπότε η Ευρώπη χρειάζεται ανθρώπους που ε, πολλά ε, πρέπει να έχουν να κάνουν με τους αλγόριθμους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερους ε, ε, ικανούς να διαβάσουν αλγόριθμους όχι μόνο στον αρμόδιο τομέα, αλλά και στο επίπεδο των ε, νομοθετών, των ρυθμιστών. Αυτή τη στιγμή, εάν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται είναι προσχεδιασμένοι, ίσως οδεύουμε προς ένα νέο συστημικό κίνδυνο, τον οποίο ακόμη δεν συνειδητοποιούμε καν. Είναι λοιπόν μια σημαντική σύσταση και αυτή. Ε, θα παραμείνω σε αυτά, Πρόεδρε, για την ώρα και ευχαρίστω να ακούσω τι παρατηρήσει των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ο κύριος Χέις από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την Κόρα για την έκθεσή της και τον τρόπο με τον οποίο ε, έδειξε διαλεκτικότητα στις συζητήσεις με τους συναδέλφους Κιώδης για να συνταχθεί η έκθεση αυτή. Απλώς μια σειρά από παρατηρήσεις σήμερα εάν μου επιτρέπετε. Η έκθεση είναι ακριβής, διεξοδική και πραγματικά χτυπάει διάνα στο στόχο. Διότι πολύ συχνά στις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας ξεφεύγουμε από το θέμα. Εδώ όμω αυτή η έκθεση πρωτοφανώ παραμένει στο κέντρο της προσοχής του, του σημείου που μας ενδιαφέρει να στρέψουμε την προσοχή μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό επίση γιατί αποστέλει ένα σαφέ μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ενθαρρύνει αυτά που εμεί ω Επιτροπή θα θέλαμε να κάνουν τα κράτη-μέλη. Να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κάνουν τα κράτη-μέλη και για τη φορολογική βάση και για το σχετικό περιβάλλον. Νομίζω είναι σημαντικό όλοι οι συνάδελφοι και όλε οι ομάδε να συνενέσουν. κάποιε παρατηρήσει για το περιεχόμενο τη έκθεση. Νομίζω ότι σαφώς πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και ε, το βασικό περιεχόμενο είναι πολύ θετικό. Καλωσορίζουμε τις συστάσεις που βάζουν την Ευρώπη σε μια τροχιά για διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών με την αξιοποίηση της FinTech, αλλά έχοντας υπόψη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών, που τα ανέφερε και η Διακόρα. Είναι λοιπόν ε, κάτι που προκύπτει με σαφήνεια την έκθεση αυτή. Εμεί ω θεσμικά όργανα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, να διευκολύνουμε μία βάση ε, ε, ανθούσα της FinTech, αλλά δίνοντα τα απαραίτητα εργαλεία στα κρατη για να πετύχουν και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών ταυτόχρονα. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε μια εύρωστη βάση FinTech σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό επίση πρέπει η διαδικασία που καταρτίζεται την έκθεση να μην λαμβάνει υπόψη μόνο τι πληρωμέ η FinTech έχει να κάνει κυρίω με υπηρεσίε πληρωμών, αλλά σωστά επικεντρώνεται και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, είναι ένα βασικό συστατικό τη έκθεση, καθώ και ε, του κινδύνου που μπορεί να, προκαλεί, να αποτύχουν από τα συστήματα πληροφορική. Πολύ σωστά τονίζονται και αυτά στην έκθεση από την εισηγήτρια. Ε, κάποια σχόλια και προτάσει για τη βελτίωση τη έκθεση θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε περισσότερο μία ε, επικέντρωση στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα περισσότερο, δηλαδή στο σχετικό τμήμα της έκθεσης. Δεν υπάρχει λόγος να ε, συμπεριλάβουμε τις νέες εξελίξεις της FinTech και αν ε, προχωράμε με, πηγαίνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Δηλαδή η χρηματοπιστωτική, σταθερότητα τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει ως προτεραιότητα αυτού του σώματος. Θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό καθώς προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε το νέο πεδίο της FinTech. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια ευθυγράμμιση και ενδυνάμωση όλων των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, στηρίζουν την χρηματοστατική σταθερότητα και σε περίπλοκες καταστάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις περιπτώσεις συστημικής ε, διαταραχής που μπορεί να προκύψει και όχι μόνο τις ανάγκες της αγοράς. Θα πρέπει η FinTech να γίνει ένα μέσο που θα επιτρέπει την ενίσχυση της νομισματικής ένωσης, όχι την ε, απλή της επίτευξη. Δηλαδή, να προωθήσουμε τους μέχρι τώρα κοινούς μας στόχους. Και μια τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε, χρήσιμο θα ήταν και η ε, Σούρτεκ να ληφθεί υπόψη ε, για τη συνολική προστασία των ε, επιχειρήσεων, διότι βλέπουμε να έχει διπλασιαστεί η παρουσία των ανώφιων εταιριών Πρέπει αυτό το νέο δυναμικό να καταγραφεί και στην έκθεση. Η Σούρτεκ δεν έχει αναπτυχθεί όπως και η Φίντεκ. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συμπεριληφθούν σε μια κοινή βάση. Καλωσορίζω λοιπόν την έκθεση και ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια για τη δουλειά τη, την αφοσίωσή τη, τη συζήτηση με όλου εμά του κοιόδη και θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε για ενδεχομένε αλλαγέ για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε, ο κύριος Ιβαν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον, την εισηγήτρια για την θαραλέα και περίπλοκη αυτή η έκθεση γιατί προσεγγίζει ένα νέο θέμα, ένα νέο τομέα, έναν κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται. Υπάρχουν πολύ σοβαρές αλλαγές που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το τι θα έχει συμβεί σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο όπως σήμερα το πώς θα πρέπει να φανταστούμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για ένα θέμα το οποίο αλλάζει συνέχεια. Μίλησα με σχετικές εταιρείε και όλα τους τα σχέδια δεν πάνε παραπέρα από ένα εξάμεινο. Δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα γίνει πέρα από αυτό τον χρονικό ορίζοντα. Γι' αυτό είναι τόσο φιλόδοξη αυτή η έκθεση. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτα απ' όλα, να ενθαρρύνουμε τα κέντρα εκείνα χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας που φαίνεται ότι λειτουργούν σε Βρετανία, ΗΠΑ, Ασία και Ολλανδία. Τα κέντρα αυτά λοιπόν να ξεπηδήσουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και να είναι σε επαφή. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε σε αυτές ε, μικρές εταιρείες ε, που μπαίνουν σε αυτή την αγορά να μην μπλοκαριστούν από τις τράπεζες. Η αντίδραση των τραπεζών μέχρι στιγμής ήταν ε, πολύ συντηρητική. Δεν θέλουν, ε, δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες και κάνουν δύσκολη την ζωή των εταιριών αυτών. αυτές ε, αγοράζονται από τις τράπεζες, ε, γίνονται τμήμα τραπεζών και χάνουν το καινοτόμο πνεύμα τους και την δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των τραπεζών και των εταιριών αυτών και των καταναλωτών για να υπάρχει μια ροή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτρέψουμε εναρμονισμένη εξέλιξη του τομέα αυτού για όλους συμμετέχοντες στην αγορά. Συζητήσαμε την φοροδιαφυγή και την καταπολέμησή της και ξέρετε πόσο σημαντικές είναι οι τράπεζες στο να μετακινούν μεγάλα ποσά σε offshore και αλλού. Είναι σημαντικό λοιπόν. Οι τεχνολογίες όπως το blockchain ή τα εικονικά νομίσματα να ρυθμιστούν και να υπάρχει διαφάνεια έτσι ώστε να μην γίνει η τεχνολογία αυτή αρνητική για τις ευρωπαϊκές κεφαλαία χώρες. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε νέους κανονισμούς ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους που υπάρχουν ήδη για τι κεφάλαια αγορές στην Ευρώπη. Μπορούσαμε να έχουμε κάποιες άλλαγες του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για να προσαρμοστούμε στην χρηματοπιστωτική τεχνολογία. Πρέπει να σκεφτούμε και τους ευπαθείς πελάτες. Να σκεφτούμε τρόπους, ε, π.χ. τα άτομα με αναπηρία άτομα τα οποία ανήκουν σε λιγότερο ευνοημένες ε, κατηγορίες ή κατοικούν σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές να έχουν πρόσβαση. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες. Δεν θα επιμείνω, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες ε, σε κάθε παράγραφο και θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ την εισηγήτρια και είμαι σίγουρο ότι θα είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ποιο είναι εδώ? Η Μπάρμπαρα Κάπελ. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω πάρα πολύ να συγχαρώ την εισηγήτρια και θα έχουμε ε, πολύ καλή συνεργασία. Πρόκειται για ένα πολύ, μια πολύ συμπαγή ε, και καλά στοχευμένη πρόταση ε, και ο στόχος μας, όπως είπατε, είναι να βρούμε μια καλή λύση, να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς για αυτό το νέο πεδίο για το, για το Κοινοβούλιο. Θέλουμε να δώσουμε ένα πλαίσιο σε όλα αυτά, κάτι που είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο. Και έρχομαι και στο πρώτο σημείο, ήδη τον ορισμό ε, του πλαισίου ε, του FinTech. Δεν είναι... Ε, μάλλον υπάρχουν κάποια προβλήματα, γιατί λέμε ότι θα πρέπει το FinTech να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, με άλλες διαπαφές. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως και η κόρα, να προωθήσουμε και για τη βιομηχανία και για την τομέα των υπηρεσιών μια σωστή λύση. Επίσης, ότι θα τα ελεγχόμενα πειράματα πάλι στους ορισμούς ε, έχω καταθέσει σχετικές ε, τροπολογίες. Υπάρχουν κάποια πειράματα που γίνονται στη Σιγκαπούρη, στην Αυστραλία. Πώς ορίζουμε το FinTech Μία τράπεζα χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε. Θα στηρίξουμε την Κομισιόν. Ε, υπάρχει το σχέδιο δράσης ε, FinTech που θα παρουσιάσει και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε σημαντικά στοιχεία. Και ένα τρίτο σημείο για τους γενικούς ορισμούς. Ε, τα πειράματα με το εικονικό ευρώ ήμουν σκιώδης εισηγήτρια στην έκθεση για τα εικονικά νομίσματα και τότε είχαμε πει ότι δεν υπάρχει ένα, αλλά αναρρύθμιτα εικονικά νομίσματα. Και σε αυτό το σχέδιο εκθέσει, θα πρέπει σας να πούμε ότι καλό θα ήταν η ΕΚΤ να έχει περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες για τα εικονικά νομίσματα. Υπάρχουν πολλά εικονικά νομίσματα. Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερες εθνικές τράπεζες. Ας εκμεταλλευτούμε τα διάφορα που υπάρχουν. Δεν ξέρω, θα δούμε τι έχει να πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο σχέδιο δράση ε, για την κυβερνοασφάλεια, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για blockchain, για νέε αλυσίδε. Η ασφάλεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και ανταλλαγή μεταξύ των ευκαιρών αρχών είναι κάτι που πρέπει να το εξασφαλίσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ασφαλείς ανταλλαγές, διαλειτουργικότητα επίσης ε, και οι τυποποιημένες ε, ε, API, Πρόσβαση επενδυτών και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με πολλούς άλλους τομείς και μας ενδιαφέρει και εδώ και στο θέμα της FinTech είναι πάρα πολύ σημαντικό και τέλος δεξιότητες είπε και η κόρα ότι για το FinTech χρειάζεται νέο πρόγραμμα σπουδών ώστε οι νέοι αλλά και αυτοί που ήδη βρίσκονται στο χώρο εργασίας να μπορούν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στο Catch the Δεν βλέπω κανένα ζητάει το λόγο. Α, είναι και η Επιτροπή εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω και εγώ να πω από την άποψη της τεχνολογίας, ε, η τεχνολογία αφορά όλο το χρηματοοικονομικό τομέα, από τις συνοφείς εταιρείε ακόμη μέχρι και τους ε, ε, καθιερωμένους τραπεζικούς φορείς το σχέδιο έκθεση είναι πάρα πολύ σφαιρικό στην προσέγγιση του. Κοιτάζει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν και να συγχαρώ την εισηγήτρια για την κάλυψη όλων αυτών των θεμάτων. Διότι πραγματικά βλέπουμε εκθέσεις ε, που, για την FinTech που ε, πλατιάζουν σε σελίδε επί σελίδων, εδώ βλέπουμε μια πολύ συνοπτική έκθεση που καταφέρνει να συνδυάσει τόσο πολλά διαφορετικά στοιχεία. Υπάρχουν πολλέ εκκλήσει για δράση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τι Ευρωπαϊκέ Εποπτικέ Αρχέ στην έκθεση και του εθνικού επόπτε. Πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο αυτό, διότι δεν υπάρχει ένας μόνος θεσμός που από μόνος του μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Οι ρυθμιστές, ο ίδιος ο κλάδος, όλοι πρέπει να δράσουν. Να δράσουν για να ε, εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίνει η καινοτομία. Επίσης, η διατομεακή προσέγγιση που δεν μπορεί να είναι μόνο χρηματοοικονομική αλλά και η πολιτική για τα δεδομένα του ανταγωνισμού, την έρευνα και ανάπτυξη, όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν. Έτσι το βλέπουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι σκοπεύουμε να χειριστούμε το όλο θέμα. Και είναι πολύ πραγματικά ε, πρόσφορο, διότι μπορεί να πετύχει αποτελέσματα που να είναι χρήσιμα για τους ίδιους τους πολίτες τελικά. Και υπάρχει και μια έκκληση για την τεχνολογική ουδετερότητα στην έκθεση. Πραγματικά αυτό γίνεται μια δυσκολία στην πράξη, διότι η ρύθμιση ε, ε, de facto αντικατοπτρίζει την κατάσταση των πραγμάτων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αντικατοπτρίζει και φωτογραφίζει την πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον. Εάν μπορούσαμε, θα γινόταν και στην νομοθεσία η πρόβλεψη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να είμαστε προετοιμασμένοι για όλε τι μελλοντικέ εξελίξει. Είναι μια δυσκολία αυτή. Σημειώνουμε ωστόσο την ε, ε, έκκληση για ε, ισοτιμότερου κανόνε του παιχνιδιού και για την αναλογικότητα. Αυτά τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν και το να χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση που να υπολογίζει και τον κίνδυνο σωστά, δηλαδή ίδιες δραστηριότητες, ε, ίδιοι κίνδυνοι, ε, ναι, είναι σωστή προσέγγιση, δηλαδή ε, συνδυάζεται με την αναλογικότητα. Και έκκληση για μια πολιτική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια, την προστασία Ναι, είναι σωστό αυτό. Αν πρέπει να επικεντρώσουμε σε κάτι την προσοχή μας, αυτό είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σημειώνουμε και μας ενδιαφέρει πραγματικά ιδιαίτερα η έκκληση για νέες τεχνολογικές λύσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στα κάτι μέλη, πρέπει να αξιοποιηθούν στον κλάδο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι βέβαια όλα αυτά γίνονται μέσα στο σωστό πλαίσιο συμμόρφωσης με την νομοθεσία και χρειάζεται και αποσαφήνιση από τις ευρωπαϊκές ε, εποπτικές αρχές που την χρειάζονται τη σαφήνεια. Στο σωστό περιβάλλον Περαιτέρω σημεία που μας απασχόλησαν στην έκθεση η ανάγκη για τη διαλογικότητα τα συστήματα να εφαρμόζονται σωστά, να υπάρχουν οι ανάλογες δεξιότητες, όχι μόνο ε, από την άποψη του ίδιου του κλάδου, αλλά και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, για τους επόπτες και τον κλάδο των εποπτών, ναι, τίνω να συμπαράνω ότι ως αποτέλεσμα των χρηματοοικονομικών τεχνολογικών καινοτομιών τα οικονομικά πλέον δεν έχουν να κάνουν μόνο με το χρήμα, αλλά με την τεχνολογία και τα δεδομένα. Και οι σχετικές πολιτικές θα πρέπει αυτό να το αντικατοπτρίσουν. Ανυπομονώ. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ήρθε και η Μαρίζα Ματίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, το συγγνώμη. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Θα ήθελα να υποφεληθώ για να κάνω κάποια σχόλια και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της πρώτα απ' όλα. Έχουμε σαφώς διαφορετικές προεπτικές για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό τα δικά μου τα σχόλια έχουν περισσότερο να κάνουν με αυτές τις αποκλήσεις της απόψης μας, περισσότερο από, τα, από σημεία, με τα σημεία στα οποία συμφωνούμε. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την έκθεση αυτή Η προσέγγιση στην έκθεση λοιπόν αυτή δίνει την εντύπωση ότι τα χρηματοποστατικά ιδρύματα περισσότερο αναζητούν την ε, ε, ευζοία των καταναλωτών και όχι το κέρδος τους. Αυτό κάπως μας ανησυχεί. Ενώ βλέπουμε να υπάρχει διαρκής και συστηματική απορρίθμιση των τραπεζικών ε, συστημάτων. Όπως χαίρει καλά η συγγήτρια, για μα η ανάπτυξη πρέπει να είναι συμμετοχική. Η τη της απασχόλησης, καταπολέμηση των ανισοτήτων. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της στρατηγικής που επιδιώκουμε. Όχι ανταγωνιστικότητα, που φαίνεται να είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εκθέση αυτής και υπό αυτή την έννοια για συμμετοχικότερη ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει και αποτελεσματικότερη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ρυθμισή του οι προτάσεις που υποβάλλονται βάζουν σε δεύτερη θέση αυτή την προτεραιότητα. Εξορισμού η FinTech δεν παρέχει καλύτερη χρηματοδότηση ή καλύτερη παροχή υπηρεσιών, ούτε καλύτερη ρύθμιση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται να εργαστούμε στο πλαίσιο της πρότασης αυτής της ΕΚΟΝ, επεδιώκοντας αυτήν την εγγύηση, αυτή την προστασία. Δηλαδή θέλουμε ρύθμιση, θέλουμε καλύτερη χρηματοοικονομική δραστηριότητα, όχι όμως με περίπλοκα προϊόντα ή με την κατανόηση των τεχνολογικών λύσεων, λες και πρόκειται για ουδέτερες τεχνολογικές λύσεις. Χρειάζεται, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι οι διάφορες τεχνολογικές λύσεις προκαλούν διαφορετικά ρυθμιστικά προβλήματα και δυσκολίες, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στην έκθεση αυτή να εμβαθύνουμε, να εμβαθύνουμε στους κινδύνους που σχετίζονται με την αυξανόμενη επιρροή της τεχνολογίας στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Αυτό είναι σαφές. Η δική μου πρόταση θα ακολουθήσει την κατεύθυνση της καλύτερης χρηματοοικονομικής ρύθμισης και τη μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή. Και αυτό βεβαίως θα έχει να κάνει με την απέτηση συγκεκριμένων και σαφών προϋποθέσεων με μια πολύ οριοθετημένη ρύθμιση. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονό ότι, όπω είπα, η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Άρα η ρύθμιση δεν μπορεί να είναι ουδέτερη σε σχέση με την τεχνολογία. Επίσης, οι τεχνολογικέ λύσεις από κάποιου ελέγχονται και πολλές φορές η τάση είναι να ε, εποφελούνται αυτοί οι οποίοι τις ε, κατασκεύασαν, τις επινόησαν το ανθρώπινο «ον» έχει ευθύνε σε πολλού τομεί, σε πολλές διαφορετικές σφαίρες. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε η έκθεση να επιμείνει λίγο παραπάνω. Και η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ε, επιμείνουμε στην προστασία του καταναλωτή και του επενδυτή. Στην πρόταση, όπω υποβάλλεται, υπάρχει απλώς μία παράγραφο σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή και του επενδυτή δεν νομίζω ότι φταίει ο περιορισμό ε, στου χαρακτήρε που προβλέπονται για τη σύνταξη τη έκθεση. Νομίζω ότι είναι επιλογή τη εισηγήτρια. Εκεί λοιπόν η διάσταση αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερη προσοχή στο πλαίσιο τη ε, διόγκωση του τομέα αυτού της fintech σε αυτήν λοιπόν την ε, κατεύθυνση ε, θα υποβάλω τις τροπολογίες μου. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη και πάλι για την καθυστέρηση. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο κύριος Ρέιμον Τόιπας. Θέλετε το λόγο? Όχι, ωραία, εισηγήτρια. Τελευταίες παρατηρήσεις. Άντε, ευχαριστώ. Επειδή έφτασα πολύ αργά. Λοιπόν, Ευγνωμονώ την κόρα για την έκθεση. Είναι πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε. Πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Μου αρέσει. Μου αρέσει η θετική της προσέγγιση. Θα πρέπει λίγο να τα συζητήσουμε βέβαια. Πώς θα βολέψουμε το να μην υπάρχει απορρίθμιση με τις νέες τεχνολογικές λύσεις. Ε, πώς θα λάβουμε υπόψη νέες τεχνολογικές λύσεις και τι θα κάνουμε με την προστασία δεδομένων, τις ασφαλιστικές εταιρείες, το αν θα πολλούνται ασφαλείς, ασφαλείς σε όσους έχουν ανάγκη από προστασία, φροντίδα, πώς όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αγορά. Και θα δούμε με την εξέλιξη των συνομιλιών μας πώς θα προχωρήσουν όλες αυτές οι ιδέες. Ευχαριστούμε και τώρα η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους Κιώδης για... και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεισφορά τους, για τα ευγενικά τους σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και να πω ότι μαζί νομίζω μπορούμε να επηρεάσουμε το μέλλον της FinTech ε, ούτως ή άλλως είναι κάτι που συμβαίνει. Εάν το εκμεταλλευτούμε, ίσως να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και απασχόληση εδώ και όχι αλλού στον κόσμο. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερο διεξοδικέ συζητήσει για πολλά από τα σημεία που αναφέρατε, όπω το να επικεντρωθούμε περισσότερο στη χρηματοπροστατική σταθερότητα, αυτό που είπατε για τη χρηματοπροστατική, τη χρηματοοικονομική ε, συμπερίληψη. Επίση, να πω στη Μαρίζα, ένα από τα τρία στοιχεία που ανέφερα στην εισαγωγή μου είναι ότι ναι, θέλω να υπάρχει προστασία του καταναλωτή στο ύψιστο δυνατό επίπεδο και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Καμία πρόθεση απορρίθμιση πίσω από αυτή την πρόταση. Και αυτό συμβαδίζει με αυτό που είπατε και εσεί για την προστασία των δεδομένων. Δεν μπορεί σε μια σύντομη έκθεση να αυτή να αναφερθούν όλα, όμω ευχαρίστω να δω τις τροπολογίες των συναδέλφων, γιατί πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με συνένεση στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 7 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Εξέταση των τροπολογιών 22 Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 10 Απριλίου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κηρύξουμε την λήξη της συνεδρίασής μας. Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στις 9 Μαρτίου στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Λήξης.